Αγαπητές και αγαπητοί συνάδελφοι, κυρίες και κύριοι, επιτρέψτε μου να σας καλωσορίσω καταρχήν εκ μέρους της Επιτροπής Ανάπτυξης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σε αυτήν την διακοινοβουλευτική σύσκεψη με τα Εθνικά Κοινοβούλια όσον αφορά την συνοχή των πολιτικών ανάπτυξης και τον συντονισμό των δωρητών Θέμα το οποίο θα συζητήσουμε με σκοπό την ενίσχυση τη συνεργασία μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και των Εθνικών Κοινοβουλίων. Λέγομαι Εύα Ζολή, είμαι πρόεδρο τη Επιτροπή Ανάπτυξη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Για μένα αποτελεί η τιμή να υποδέχομαι σήμερα εδώ τι αντιπροσωπείε των Εθνικών Κοινοβουλίων. Η συνεργασία μεταξύ επιτροπών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και των ε, αντιστοίχων επιτροπών των Εθνικών Κοινοβουλίων αποτελεί σημαντική επιταγή στον καιρό μας για να γνωριστούμε μεταξύ μας καλύτερα και να επιτύχουμε συνοχή ο καθένα στην Επιτροπή του με γνώμονα βεβαίω την αυξημένη αποτελεσματικότητα και απόδοση. Με λιγότερα να κάνουμε δηλαδή περισσότερα. Γι' αυτόν τον λόγο το θέμα το σημερινό μου φαίνεται ενδιαφέρον και χρήσιμο. Ελπίζω ότι η σημερινή συζήτηση θα συμβάλλει στην ανάδειξη των δυνατοτήτων της συνεργασίας μας και ενδεχομένω να οδηγήσει σε περισσότερη διαβούλευση και συνεννόηση καθώς και συντονισμό μεταξύ των εθνικών πολιτικών και της πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης στον τομέα της συνοχής και του συντονισμού των πολιτικών ανάπτυξης. Όπως ε, προβλέπετε και στην ημερήσια διάταξη, η σημερινή μας σύσκεψη, η σημερινή μας συνεδρίαση ε, θα ξεκινήσει υπό την προεδρία του κυρίου Γκέρενς. Θα μιλήσουμε για την συνοχή των πολιτικών για την ανάπτυξη εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτό είναι το πρώτο μέρος. Κατά τη διάρκεια αυτού τα Εθνικά Κοινοβούλια θα καταθέσουν παραδείγματα καλών πρακτικών από τη χώρα τους και το οποίο θεωρώ ότι θα συμβάλλει σε μια επικοδομητική μεταξύ μας συζήτηση. Στο δεύτερο μέρος, τον κύριο Κιμισελ, θα έχει ως θέμα τα εργαλεία και τα όργανα για τον περαιτέρω συντονισμό των πολιτικών ανάπτυξη εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης με γνώμονα την βελτίωση ακριβώ τη βοήθεια, τη αναπτυξιακή βοήθεια. Και θα κλείσουμε με τον κύριο Πατ Μπριν, πρόεδρο της, ε, της Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων και Εμπορίου του Ελληνικού Κοινοβουλίου και αν ο χρόνος το επιτρέψει θα ακούσουμε μια σύνοψη και από των δύο θεμάτων της σημερινής συνεδρίασης. Πριν δώσω τον λόγο στον Επίτροπο Πίλμπαξ, θα ήθελα να υπογραμμίσω ότι η συνοχή των πολιτικών ανάπτυξης δεν είναι συνοχή μεταξύ των εθνικών πολιτικών και αυτής της Ένωσης αφορά όλες τις εξωτερικές πολιτικές της Ευρωπαϊκής Ένωσης και ένα εξαιρετικό παράδειγμα είναι η Νορβηγία. Η Νορβηγία δημιούργησε ένα ταμείο το οποίο προκοδοτήθηκε πλούσια με 3 δισεκατομμύρια δολάρια για την αντιμετώπιση της ε, καταστροφής των δασών. Βεβαίω ε, νορβηγικές επιχειρήσει κατασκευάζουν ε, ένα τεραστίο φράγμα στον ε, Αμαζόνιο και συμβάλλουν και στην αποδάσωση. Βλέπετε λοιπόν ότι ότι πολλές φορές υπάρχουν ιστορικές αντιφάσεις, αυτό πρέπει να κατανοήσουμε και γι' αυτό πρέπει να κάνουμε κάτι και γι' αυτό είμαστε εδώ. Οι γερμανικές επιχειρήσεις, οι επιχειρήσεις της Αυστρίας, της Νορβηγίας, όταν δραστηριοποιούνται σε αναπτυσσόμενες χώρες πρέπει να σέβονται και εκεί το περιβάλλον και όχι μόνο στις χώρες τους. Κύριε Πίλμπαξ, έχετε το λόγο. Thank you. Uh, thank Ευχαριστώ. κύριε Πρόεδρε, αξιότιμα μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, αξιότιμα μέλη των Εθνικών Κοινοβουλίων, κυρίες και κύριοι. Είναι τιμή μου να παραβρίσκομαι σε αυτή την διακοινοβουλευτική συνάντηση, γιατί Πρόκειται για μια ευκαιρία να επανενώσουμε τις δυνάμεις μας για να αντιμετωπίσουμε αυτές τις εξελίξεις. Εσείς που υπερασπίζεστε την ανάπτυξη, τα γνωρίζετε αυτά, δεν θα κάνω μια μακρά εισαγωγή, αλλά θα ήθελα να τονίσω τρία σημαντικά ζητήματα. Το ένα είναι ότι δεν υπάρχουν ε, εξελίξεις, δεν υπάρχει ε, βιώσιμη ανάπτυξη για την ειρήνη και δεν υπάρχει ούτε ευημερία, ακόμη και αν δούμε την παγκοσμία ανάπτυξη. Γι' αυτό η αναπτυξιακή συνεργασία είναι τόσο σημαντική, γιατί παρέχει ένα βιώσιμο μέλλον για όλους μας και Υπό το πρίσμα αυτό, η σημερινή συζήτηση θα αγγίξει δύο σημαντικά ζητήματα στη σημερινή αναπτυξιακή πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Θα σας δώσω κάποια αριθμητικά στοιχεία για να καταλάβετε τις δεσμεύσεις πέρσι σε πληρωμές. Αυτό σημαίνει το 2012. Η συνολική επίσημη αναπτυξιακή βοήθεια από την Κομισιόν ήταν 9 δισεκατομμύρια ευρώ. Ένα δισεκατομμύριο είναι ανθρωπιστική βοήθεια, δηλαδή ουσιαστικά 8 δισεκατομμύρια δόθηκαν ε, μέσω της κοινότητας ε, και περίπου 50 δισεκατομμύρια ε, είχαμε από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Έτσι λοιπόν σημαίνει ότι ο συντονισμός είναι πάρα πολύ σημαντικός αν θέλουμε να πετύχουμε τα βιώσιμα αποτελέσματα και αυτό το βιώσιμο πλαίσιο αποτελεσμάτων. Από μια άλλη σκοπιά, αν δούμε αυτά τα 8 δισεκατομμύρια σε σύγκριση με τις ανάγκες της Αφρικής για την ενέργεια και τις σχετικές επενδύσεις, θα έπρεπε να φτάσουμε στα 50 δισεκατομμύρια. Και αυτό σημαίνει ότι θα πρέπει να δούμε ποιες είναι άλλες πηγές για ανάπτυξη. Ε, θα πρέπει βέβαια κάποιος να δει τους εγχώριους φόρους ε, και φυσικά αυτό εξαρτάται από τη συνοχή της αναπτυξιακής πολιτικής. Αλλά υπάρχουν και άλλα σχετικά θέματα όπου οι πολιτικές της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το εμπόριο, στη γεωργία, στην αλία με τη δική μας προσέγγιση για τα παγκόσμια ζητήματα έχουν πολύ μεγάλη επίπτωση στη δυναμική των χωρών να ακολουθήσουν αναπτυξιακά μονοπάτια. Έτσι λοιπόν η συνοχή της αναπτυξιακής πολιτικής, ακόμη και αν ακούγεται ως μια πλουστευμένη προσέγγιση, θα μπορούσε σε μεγάλο βαθμό να έχει μεγαλύτερο αντίκτυπο από τις άμεσες αναπτυξιακές ροές. Έτσι λοιπόν αυτά τα θέματα σχετίζονται πάρα πολύ με τις ε, πληρωμές ε, για την υποστήριξη των αναπτυσσόμενων χωρών, αλλά ταυτόχρονα πρέπει να κατανοήσουμε με σαφήνεια ότι αυτός ο συντονισμός μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και άλλων εταίρων, δίχως δηλαδή αυτό το συντονισμό και χωρίς τη συνοχή δεν μπορούμε να περιμένουμε ότι τα κονδύλια για την ανάπτυξη θα έχουν ε, ουσιαστική προσθεμένη αξία. Αυτό που προσπαθούμε τώρα να πετύχουμε στο συντονισμό σχετίζεται ιδιαίτερα με τον κοινό προγραμματισμό, όπως τον αποκαλούμε, joint programming. Αυτό τι σημαίνει ουσιαστικά ότι βλέπουμε το αναπτυξιακό σχέδιο των αναπτυσσόμενων χωρών, κάποιων αναπτυσσόμενων χωρών με τις πληρωμές που έχουν προβλεφθεί και προσαρμόζει στη δική σου αναπτυξιακή στρατηγική εναντί αυτού του αναπτυξιακού σχεδίου, προ αυτό το αναπτυξιακό σχέδιο και ταυτόχρονα προσπαθεί εντό τη Ευρωπαϊκή Ένωση να εργαστεί για να έχει το ίδιο πλαίσιο αποτελεσμάτων και τον ίδιο ρυθμό ανάπτυξη πολιτικά. Όλοι οι συναδελφοί μου το υποστηρίζουν αυτό. Και χτες υπήρχε μια συμφωνία να αφαιρθούν όλες οι κυρώσεις από τις σχέσεις μας με τη Βερμανία και ε, κλήθηκαν ε, οι Υπουργοί Εξωτερικών να εφαρμόσουν ένα κοινό προγραμματισμό έτσι λοιπόν αυτό σημαίνει ότι όλες οι ευρωπαϊκές χώρες το υποστηρίζουν αυτό θεωρητικά, αλλά όταν φτάνουμε στην εφαρμογή είναι διαφορετικές οι προκλήσεις, γιατί αυτό θίγει τους συνήθεις κύκλους προγραμματισμού, επίσης έχει επίπτωση στα συγκεκριμένα μοντέλα που έχουν καθιερωθεί για 50, 20, 10 χρόνια, αλλά χρειάζονται πάρα πολλές αλλαγές και νομίζω ότι είναι ζωτικό τα εθνικά κοινοβούλια να ζητούν ε, από την πολιτική συνεργασία ε, και από τους αρμόδιους για την ε, συνεργασία αυτή την απτυξιακή και από τους οργανισμούς να ακολουθήσουν αυτό το μοντέλο γιατί σε ορισμένες χώρες είδαμε ότι τα Υπουργεία της χώρας Εταίρου, το Υπουργείο Γεωργίας στο Μαλάουι παραδείγματος χάρη ε, τελικά είναι μια μονάδα που απλώς εξυπηρετεί τα project, γιατί έχουν τόσα πολλά έργα, τόσο πολλά project και οι διοικητικέ ε, ικανότητες χρησιμοποιούνται μόνο και μόνο για να παρακολουθούνται αυτά τα προγράμματα και ουσιαστικά δεν υπάρχει καμία στρατηγική συνοχή στο Υπουργείο γιατί δεν, ε, έχει, δεν έχουν απομείνει διαθέσιμοι πόροι. Έτσι λοιπόν, η άποψή μου είναι ότι κοινός προγραμματισμός δεν αποτελεί εξαίρεση αλλά τον κανόνα. Αλλά πρόκειται για κανόνε που δεν μπορούμε να επιβάλλουμε, θα πρέπει να γίνουν αποδεκτοί αυτοί οι κανόνε. Ε, σε πολιτικό επίπεδο γίνονται <coughs> αποδεκτοί, ενώ σε διοικητικό επίπεδο χρειάζεται ακόμη δουλειά. Και δεν είναι καινούργια αυτή η διαδικασία. Σε επίπεδο Ευρωπαϊκής ε, Ένωσης η ενοπτυξιακή βοήθεια του 2007 ζητούσε συμπληρωματικότητα και κατανομή της εργασίας και μετά από έξι χρόνια εξακολουθούμε να παλεύουμε για να επιτευχθούν αυτά. Όμως ε, φαίνεται πως υπάρχουν σημαντικές αλλαγές. Ε, εγώ συμμετείχα σε μια συνέντηση με την κυβέρνηση της Αιθιοπίας ε, και με όλες τις αντιπροσωπείες της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην Νορβηγία και την Νορβηγία και κάναμε μια ανάλυση για τον κοινό προγραμματισμό και φαίνεται ότι θα υλοποιηθούν αυτά και αναμένω το 2014 θα μπορούσαμε να έχουμε κοινό προγραμματισμό με την Αιτή, το Σουδάν, τη Ρουάντα, τη Γουατεμάλα, την Κάνα, την Αμίμπια και την Αίγυπτο. Κινούμαστε λοιπόν, αλλά αν ε, ε, μιλήσουμε για έναν αριθμό 150 χωρών, ε, για τη βοήθεια που θα φτάσει σε 150 χώρες, μόνο ξεκινάμε. Επομένως πρέπει να εργαστούμε έτσι και αυτός να είναι ο κανόνας. Και ιδίω αυτά είναι σημαντικά στη νέα περίοδο, δηλαδή από το 2014 έως το 2020. Γιατί αυτή είναι μία περίοδος όπου η αναπτυξιακή βοήθεια της Ευρωπαϊκής Ένωσης ε, προετοιμάζεται για τα επόμενα 7 έτη και έχουμε πραγματικά την ευκαιρία να την προετοιμάσουμε στο ρυθμό των ε, αναπτυσσόμενων των ε, χωρών εταίρων μας ε, και να έχουμε μια κοινή προσέγγιση. Γιατί είναι δύσκολο να το κάνουμε αργότερα, γιατί έχουμε δύο δημοσιονομικές αρχές, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο και να κάνουμε αλλαγές αργότερα είναι μια ιδιαίτερα βαριά διαδικασία και έτσι λοιπόν εγώ κατανοώ ότι η Κομισιόν θα πρέπει να δώσει το παράδειγμα για τον κοινό προγραμματισμό, όμως έχουμε ένα περιορισμένο χρονικό διάστημα για να το πετύχουμε αυτά. Έτσι λοιπόν θα να έκκληση σε όλους εσάς να υποστηρίξετε το κοινό προγραμματισμό αλλά <coughs> και να ζητήσετε από τους συναδέλφους σας στις κυβερνήσεις και από τους αναπτυξιακούς οργανισμούς να τους ρωτήσετε πώς προχωρά αυτό το έργο. Και επαναλαμβάνω, θα πρέπει να είναι ο κανόνα και όχι η εξαίρεση. Και σήμερα εξακολουθούμε να εργαζόμαστε επί εξαιρετικών καταστάσεων και δεν βλέπω καμία δικαιολογία γι' αυτό. Γιατί αν ε, δεν εργαστούμε στο πλαίσιο του κοινού προγραμματισμού, τότε βασικά θα χαθεί ένα τμήμα της αξίας ε, των κονδυλίων. Έχουν γίνει κάποιοι υπολογισμοί, αλλά αυτό βασικά σημαίνει ότι αν δουλέψουμε μέσω κοινού προγραμματισμού, τότε αυξάνουμε τη βοήθεια, ε, βελτιώνεται κατά 6 δις. Θα κερδίσουμε δηλαδή αυτά τα 6 δισεκατομμύρια. Υπάρχουν κάποια θέματα ιδιαίτερα σχετικά με αυτό. Δεν είναι στη σημερινή ημερήσια διάταξη, αλλά μια ανησυχητή τάση είναι η αναπτυξική βοήθεια από τις αρχής. Γιατί Πέρσι δεν ήταν πολύ καλό το έτος για την επίσημη αναπτυξιακή βοήθεια. Ήταν μεικτά κάπως τα συναισθήματα για πέρσι, μικτές οι εντυπώσεις, γιατί υπήρχαν κάποιες χώρες όπου είδαμε κάποιες ε, βελτιώσεις. Ε, φαίνεται να ήταν αμυκτά τα αποτελέσματα. Πέρσι όμως ε, οι στατιστικές ε, για φέτος της αναπτυξιακής βοήθεια είναι καταστροφικές. Από τη σκοπιά ότι καταρχήν ε, από το από το 0,42 πέσαμε και αυτό είναι στο 0,39 του ακαθάριστου χώρου προϊόντος ε, και αυτό είναι καταστροφικό. Ε, γιατί δεν υπάρχει εξαίρεση για τα κράτη-μέλη. Είχαν πει ότι θα δεσμευτούν για 0,7. Αλλά όταν δούμε τι συμβαίνει στην πράξη δεν ισχύει κάτι τέτοιο. Και αν ε, δούμε τι συνέβη με το ποσό που δόθηκε στο τελευταίο πακέτο διάσωσης ε, για ένα κράτος μέλος ήταν 10 δισεκατομμύρια. Και ενώ πέρσι είχαμε δαπανίσει 9 δισεκατομμύρια και για την ανθρωπιστική βοήθεια. Έτσι λοιπόν θέλω να απευθύνω έκκληση στι κυβερνήσει να σεβαστούν τι υποσχέσει του. Όμω δεν πρόκειται για φιλανθρωπία. Είναι επένδυση για περισσότερη ασφάλεια. Γιατί αν δεν το κάνουμε αυτό τότε θα έχουμε περισσότερε στρατιωτικέ δαπάνε. και ε, αν υπάρχει κρίση θα πρέπει να δώσουμε περισσότερη ανθρωπιστική βοήθεια για να υποστηρίξουμε του ανθρώπου στην κρίση. Η ανθρωπιστική βοήθεια δεν είναι απάντηση απλώς ε, αποτελεί μια γέφυρα για την κανονική ζωή, αλλά πώς θα ανακτήσουμε την ε, κανονική ζωή. Και αν δούμε τις προκλήσεις ε, που έχουμε ενώπιόν μας, όπως η Συρία και η νοικοδόμηση του Μαλή και το Σαχέλ, χρειαζόμαστε πάρα πολλά να κάνουμε εκεί και στο κέρας της Αφρικής δεν ε, βλέπω να μπορούμε να ε, παράσχουμε ασφάλεια και ευημερία για τους Ευρωπαίους πολίτες ε, και πραγματικά μας ανησυχεί πάρα πολύ το τι συμβαίνει σήμερα. Όπως σας είπα δεν είναι στη σημερινή ημερησία διάταξη, αλλά δεν μπορούμε να αποφύγουμε να μιλήσουμε για τον συντονισμό της βοήθειας. Αν υπαναχωρούμε ε, και δεν σεβόμαστε τις υποσχέσεις που έχουμε δώσει στις χώρες εταίρους, αλλά ούτε επιδιώκουμε να πετύχουμε τα συμφέροντα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ως ε, πλαίσιο υπάρχει μια συμφωνία για την περίοδο 2014-2020 και ε, αυτή τη στιγμή έχουμε περίπου στο 60% και δεσμεύονται μόνο οι εθνικοί προπολογισμοί. Έτσι λοιπόν η δυνατότητα ε, να επαναπροσδιορίσουμε το πώς λειτουργεί ο προπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης και να μπουν περισσότερα χρήματα εκεί είναι περιορισμένη δυνατότητα. Αλλά πιστεύω ότι οι εθνικοί προπολογισμοί πρέπει να αυξηθούν και είναι ζωτικό και για τα δικά μας συμφέροντα. Τώρα, η συνοχή της αναπτυξιακής πολιτικής. Νομίζω ότι η συνοχή της αναπτυξιακής πολιτικής είναι κάτι το οποίο το έχουμε υπερτονίσει ως Ευρωπαϊκή Ένωση και όλοι μας προσπαθούμε να την προωθήσουμε και σωστό είναι. Αλλά αν δούμε τι έχουμε αλλάξει στην πραγματικότητα, πρόκειται μόνο για κάποια στοιχεία τα οποία έχουν αλλάξει ουσιαστικά. Είμαι πολύ περηφανός ε, για την οδηγία διαφάνειας για τις εκτοριστικές βιομηχανίες ε, που κατέθεσε ο Μισελ Μπαρνιέ και ευθύθηκε από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Γιατί η αναπτυξική βοήθεια και μόνο δεν αρκεί. Είναι σαφές αυτό. Ταυτόχρονα λέμε ναι, οι αναπτυσσόμενες χώρες έχουν ιδίους σπόρους και θα μπορούσαν να εκμεταλλευτούν περισσότερο τους σπόρους αυτούς. Όμως δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι αυτές οι χώρες είναι μικρές, ευάλωτες και διαπραγματεύονται με πολυεθνικές που έχουν όλες τις εξουσίες στη διαπραγμάτευση. Έτσι λοιπόν τελικά οι συμφωνίες για τις χώρες αυτές δεν είναι βέλτιστες και είναι κρίμα ότι μέχρι τώρα δεν υπήρχε ουσιαστικά καμία ενημέρωση ένα project για το τι παίρνει κάθε χώρα σε αυτό και υπήρξε μεγάλη ε, αυτό και εγώ νομίζω ότι η διαφάνεια είναι το πρώτο βήμα προς την ευημερία. Πιστεύω λοιπόν ότι είναι ένα καλό παράδειγμα όπου θα μπορούσαμε εμείς να δείξουμε ότι έχει νόημα η συνοχή της αναπτυξιακής πολιτικής μας. Με αυτό σχετίζεται ένα θέμα με την ξυλία. Τώρα έχουμε ένα κανονισμό που ε, σύμφωνα με το νομίο μπορεί να εισάγει η Ευρωπαϊκή Ένωση ε, μόνο ξύλια που έχει κοπεί νομίμως και εφαρμόζουμε το FLEGT για να οθήσουμε και τις χώρες εταίρους προς την αηφόρο διαχείριση των δασών. Έχουμε πολύ δρόμο μπροστά μα αλλά όλο και περισσότερες χώρε εντάσσονται σε αυτό. Ολοκληρώσαμε τι διαπραγματεύσει με την Ενδονησία, το χάρη. Και αν ακολουθήσουμε αυτή την προσέγγιση, όλοι θα κερδίσουν. Γιατί μιλάμε πραγματικά για η φόρο διαχείριση των δασών και ταυτόχρονα ε, κόβουμε ένα μεγάλο αριθμό των παράνομων ροών. Έχει Βέβαια, αυτό που έχει σημασία είναι τα αποτελέσματα, αλλά ε, αυτό σχετίζεται με την ε, καταπολέμηση της φοροαποφυγής. Γιατί εδώ θέλουμε να έχουμε διαφάνεια στις χρηματοοικονομικές ροές. Πολλές φορές βλέπω ότι είναι πολύ δύσκολη κατάσταση όταν οι συνάδελφοι για τις χώρες λένε υπάρχουν έχουν ε, κάποια χρήματα που ουσιαστικά τα κλέβουν από τους πολίτες αυτής της χώρας και πηγαίνουν προς ε, φορολογικούς, όχι προς φορολογικούς παραδείσους, αλλά εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης και προσπαθούν να ανακτήσουν αυτά τα ποσά και δεν υπάρχει τέτοια δυνατότητα. Όμως εγώ νομίζω ότι θα πρέπει να αγωνιστούμε για τη διαφάνεια και την λογοδοσία ε, για αυτές τις πληρωμές, ε, όχι μόνο παγκοσμίω, αλλά και εντό της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπου θα μπορούσαμε να σημειώσουμε σημαντική βελτίωση σε αυτά τα θέματα, γιατί είναι δύσκολο τελικά να περασπίσουμε όλες τις απαιτήσει για διαφάνεια και την καταπολέμηση της διαφθοράς, αν έχουμε κάποιες γκρίζες ζώνες όπου μπορούν να παρεκκλίνουν τα χρήματα από αυτές τις χώρες και κατόπιν δεν μπορεί να υπάρχει πρόσβαση σε αυτές τις γκρίζες ζώνες. Έχουμε δει λοιπόν ε, ότι και τα έσοδα, ε, με αυτόν τον τρόπο και τα αφορολογικά μας έσοδα θα αυξηθούν. Όμως, επίσης, ήμουν ιδιαίτερα ικανοποιημένος από το εξή ότι ο κύριος Τσόλος, ο συνάδελφος που είναι αρμόδιος για τη Γεωργία, δημοσίευσε να ότι ε, θα καταργήσει όλες τις εξαγωγικές πιστώσεις για τα γεωργικά προϊόντα. Είναι σημαντικό να θέσουμε ένα τέλος ε, και σε αυτό και επίσης το εμπόριο έχουμε σημειώσει σημαντικά επιτεύγματα αλλά και εκεί υπάρχει περιθώριο βελτιώσεων και ελπίζω ότι η συνέχιση των διαπραγματεύσεων για τις ε, συμφωνίες εταιρικής σχέσης θα μπορούσε να βελτιωθούν. Θα έλεγα λοιπόν συνολικά ότι η προσέγγιση μας για τη συνοχή της αναπτυξιακής πολιτικής έχει πάρα πολλά θετικά αποτελέσματα για τις χώρες ε, ε, εταίρους μας. Έχουμε πετύχει πολλά, αλλά θα μπορούσαμε να κάνουμε πολλά περισσότερα, γιατί εγώ πιστεύω ότι εμείς είμαστε σε ηγετική θέση στη συνοχή της αναπτυξιακής πολιτικής, αλλά θα πρέπει να συνεχίσουμε να προωθούμε αυτή την προσέγγιση και φυσικά καλό και τα μέλη των κοινοβουλίων να μας υποστηρίξουν σε αυτό. Γιατί πολλές φορές φαίνεται σαν να θίγονται τα συμφέροντα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά αυτό είναι λάθος. Δεν ισχύει γιατί όσο περισσότερη διαφάνεια έχουμε, θα έχουμε και περισσότερη ισότητα στο εμπόριο και περισσότερη συνοχή μεταξύ των διάφορων πολιτικών. Όλα αυτά ενδυναμώνουν την Ευρωπαϊκή Ένωση και θα έχουμε περισσότερο εισόδημα και για μας. Και νομίζω ότι αυτό δεν θα πρέπει να το δούμε από μια στενή οπτική μια συγκεκριμένη ομάδα ε, λόμπι, αλλά θα πρέπει να δούμε πώς ωφελούνται οι πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης από αυτό, από τη συνοχή της αναπτυξιακής πολιτικής. Έτσι λοιπόν, εύχομαι κάθε επιτυχία για τη σημερινή συνεδρίαση, για τη συνοχή της αναπτυξιακής πολιτικής. Ε, θα παρουσιάσουμε και μία έκθεση το φθινόπωρο. Θα προσπαθήσουμε να δείξουμε τα θετικά που θα έχουμε πετύχει και τις προκλήσεις που πρέπει να αντιμετωπίσουμε. Και για το κοινό προγραμματισμό επίσης ε, θα ενημερώσω το Κοινοβούλιο τον Οκτώβριο ότι θα έχουμε πετύχει σε εκείνο το στάδιο γιατί θα είναι πραγματικά ζωτικό να έχουμε ένα σαφές follow-up ε, για ποιες χώρες μιλάμε και έχουν κοινό προγραμματισμό και που βρισκόμαστε με τις υπόλοιπες χώρες γιατί αν ε, δεν κάνουμε τουλάχιστον κοινό προγραμματισμό τότε αυτό θα είναι αδικαιολόγητο. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ και εγώ κύριε Πιμπάλξ. Θα ήθελα τώρα να ξεκινήσουμε μια συζήτηση, σύντομη ανταλλαγή απόψεων με τον ε, Επίτροπο. Σας καλώ όταν πάρνετε το λόγο να λέτε ποιοι είστε και από πού έρχεστε. Δεν έχουμε πολύ χρόνο στη διάθεσή μας, οπότε είστε λακωνικοί. Λέγομαι Κάρεν Ροτ, από τη Γερμανία είμαι από την πολιτική ομάδα των Σοσιαλδημοκρατών. Ευχαριστώ πάρα πολύ ε, για την παρουσίαση αυτή κύριε Πίμπαλξ. Όντως ε, χαίρομαι για αυτά που είπατε, χαίρομαι για αυτά που είπατε για την εφαρμογή και για το ότι τονίσατε την, τον κοινό προγραμματισμό. Αυτός πράγματι χρειάζεται ε, και νομίζω ότι... Ε, πρέπει να σας υποστηρίξουμε και τα Εθνικά Κοινοβούλια το ίδιο. Αλλά θέλω να ρωτήσω κάτι τι, για έναν τομέα που δεν είναι δική σας αρμοδιότητα βέβαια, αλλά... θα, θα ήθελα να πείτε μερικά πράγματα και για την έρευνα και για τα ε, γεωργικά θέματα και για τις εμπορικές συμφωνίες δεν θα μπορούσε να φτιαχτεί μια πολυκλαδική ομάδα τρόπων τεινά για να συζητηθούν και αυτά τα θέματα και να συντονιστούν και όλοι εκείνοι οι τομείς που έχουν επιπτώσεις γιατί όλα αυτά έχουν επιπτώσεις ένα πτυσσόμενες χώρες. Αυτή η ιδέα λοιπόν μιας πολυκλαδικής μιας, ενός πολυκλαδικού συντονισμού των επιτρόπων ίσως τα λέγαμε ούτως ώστε και η νομοθεσία και οι οδηγίες και τα λοιπά να είναι συντονισμένες Ευχαριστώ πολύ, έχετε το λόγο Έχει μικρόφωνο ο μιλητής um, first of all, Πρώτα πρώτα, κύριε Επίτροπε, θα ήθελα να σας ευχαριστήσω για όλα αυτά που μας είπατε. Βεβαίως θα πάρω και το λόγο αργότερα και συμφωνώ πολύ με αυτά που είπατε, αλλά έχω ένα ειδικό θέμα για την ασφάλεια των τροφίμων και την ασφάλεια προ, προμήθειας τροφίμων και έχουμε ένα πρόβλημα με τη βιομάζα και την ενέργεια από και τα βιοκαύσιμα ας πούμε ε, υπάρχουν στις νομοθετικές πράξεις της κοινότητας ορισμένα πράγματα τα οποία είναι αντίθετα προς την ε, ασφάλεια φοδιασμού με τρόφιμα. Θέλω να ρωτήσω, πιστεύετε ότι αυτό το θέμα δεν θα πρέπει να μελετηθεί, γιατί αυτό πιστεύουμε ότι είναι σημαντικό, γιατί ουσιαστικά τα εσωτερικά συμφέροντα της κοινότητας συγκρούονται με τα εξωτερικά και με την βοήθεια προς αναπτυσσόμενες χώρες προφανώς. I give the floor to Mr. to answer. Ο κύριος Πίμπαλξ θα απαντήσει αυτές τις δυο ερωτήσεις. Εν τω μεταξύ εσείς μπορείτε να προετοιμάσετε τις επόμενες. Ο Επίτροπος θα ήθελα να πω πρώτα πρώτα ότι όλοι μας μάλλον ότι γίνεται αξιολόγηση του αντικτύπου όλων των αποφάσεων που παίρνει το σώμα των επιτρόπων η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και όλα αυτά αναλύονται και όσον αφορά τις επιπτώσεις για την ε, αναπτυξιακή βοήθεια. Ε, δηλαδή όλοι οι επίτροποι προσπαθούν να συντονιστούν. Συγχρόνως πρέπει να εντοπίσουμε τους τομείς όπου θα μπορούσαμε να πετύχουμε τα καλύτερα αποτελέσματα. Και σε αυτό το στάδιο επικεντρώνουμε τις προσπάθειές μας σε διμερείς παφές, αν θέλετε με ορισμένους συναδέλφους. Εσείς αναφέρατε την έρευνα και άλλους τομείς όπου α, υπάρχουν Εν και άλλους μισό που θα μπορούσαμε να επηρεάσουμε τα πράγματα και ξέρω ότι ε, ασχολείστε και με τις σπάνιες ασθένειες κτλ Όντω όντως θα πρέπει να υπάρξει συντονισμός και συνοχή ανέφερα προηγούμενα τον Μισελ Μπαρνιέ ο οποίος είναι υπεύθυνο για την ε, ε, ε εσωτερική αγορά ανέφερα τον κύριο Τσόλος της Γεωργίας η κυρία Δαμανάκη είναι υπεύθυνη για την αλία και με αυτούς ήδη συντονιζόμαστε γιατί υπάρχει μεγάλη επίπτωση των πολιτικών μας στις αναπτυσσόμενες χώρες Ο, αλλά από εκεί και πέρα βεβαίως υπάρχουν και άλλοι τομείς στους οποίους πρέπει να ε, φροντίσουμε να υπάρχει συντονισμός κάνουμε συντονισμό αλλά ίσως δεν αρκεί είναι σαν το κοινό προγραμματισμό ε, θα πρέπει να δουλέψουμε παραπάνω είναι γεγονός. Είναι πολύ σημαντικό να, να λάβουμε επιπλέον δράσεις και πρωτοβουλίες αλλά δεν μπορώ να επικρίνω τους συναδέλφους επιτρόπους γιατί δεν κάνουν πράγματα παραπάνω έχουν ήδη πάρα πολλά άλλα πράγματα να κάνουν τώρα θα αναφερθώ στα βιοκάψιμα που αναφέρθηκαν στην πολιτική μας για την ενέργεια πήραμε μία πολύ σαφή απόφαση ότι δεν θα υποστηρίξουμε κανένα έργο που σχετίζεται με τα βιοκαύσιμα. Και στην εσωτερική εσωτερική νομοθεσία και η εσωτερική μας νομοθεσία για την βιωσιμότητα των βιοκαυσίμων ενισχύεται αυτή τη στιγμή. Χαίρομαι που γίνονται αυτά. Ξέρω βεβαίως ότι το ερώτημα σας σχετίζεται με τους στόχους για τα βιοκαύσιμα. Δεν είμαι αρμόδιος για τα θέματα αυτά αλλά ποια ήταν η βασική ιδέα η βασική ιδέα ήταν να προχωρήσουμε στη δεύτερη γενιά βιοκαυσίμων με απόβλητα, με κατάλοιπα και με επανεπεξεργασία των προϊόντων αυτών. Ελπίζω αυτές οι πολιτικές να προχωρήσουν γιατί υπάρχει και αντίθετη όψη, αντίθετη πλευρά που πρέπει να έχουμε υπόψη μας. Δηλαδή οι γεωτρήσεις για το πετρέλαιο και η χρήση των ορυκτών καυσίμων επηρεάζει το περιβάλλον ακόμη και αν δεν συμβαίνει στην Ευρωπαϊκή Ένωση, επηρεάζει το περιβάλλον αρνητικά εκτό της Ευρωπαϊκής Ένωση. Είναι πολύ σημαντικά αυτά τα πράγματα για την ενέργεια. Από τη μια θέλουμε λοιπόν ενεργειακή αποδοτικότητα, αυτό και τώρα κάνω μια παρένθεση εξεπλάγει θετικά για τις Ηνωμένε Πολιτείες της Αμερικής ε, γιατί στις Ηνωμένε ε, πολιτείες ορισμένα πράγματα δεν πήγαιναν καλά αλλά τα πράγματα τώρα άλλαξαν και είδα ότι άλλαξαν τα πράγματα στις Ηνωμένε Πολιτείε. Δεν ξέρω πώς το κατάφεραν και τουλάχιστον άλλαξε και η, η τακτική αυτή, η συνήθεια αυτή που κάνουν τα πάντα ψυγείο. Ε, ε, βεβαίως δεν πρέπει να αγνοούμε και την ανάπτυξη των νέων τεχνολογιών στις ε, τηλεπικοινωνίες λόγου χάρη, οι νέες τεχνολογίες οδήγησαν σε επανάσταση. Στον τομέα της ενέργειας δεν έγινε κάτι τέτοιο, αλλά θα πρέπει να επιμείνουμε στην ανάπτυξη νέων τεχνολογιών και στον τομέα της ενέργειας, διότι διαφορετικά ε, δεν θα μπορέσουμε να μειώσουμε την εξάρτησή μας από τα ορυκτά καύσιμα. Χρειαζόμαστε τις ανανεώσιμες ενέργειες, να διπλασιάσουμε την αποδοτικότητα, την ενεργειακή. Ε, χρειαζόμαστε νέες τεχνολογικές ε, λύσεις. Αν δεν τα κάνουμε όλα αυτά δεν θα μπορέσουμε να προχωρήσουμε και θα παραμείνουμε και σε μια δύσκολη δεσμενή κατάσταση όσον αφορά την ανάπτυξη των βιοκαυσίμων. Η Βραζιλία κάνει θαύματα, ε, και, αλλά ε, πρέπει να ακολουθήσουμε και εμείς. Εμείς, εν πάση περιπτώσει, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή υποστηρίζει όλες αυτές τις ιδέες πάντως. Λουί Μισελ. Κύριε Πρόεδρε, συγχαρητήρια πρώτα απ' όλα για τη σημερινή συνεδρίαση. Σπάνια έχουμε την ευκαιρία να συναντούμε τα Εθνικά Κοινοβούλια και να έχουμε και τη δυνατότητα να στείλουμε κάποια μηνύματα. Η πρόσκληση αυτή ήταν πολύ σημαντική. Πρώτον, ω προ την κατανομή εργασία. Ο Επίτροπο το είπε. Το κόστος του κατακαιρματισμού των διαδικασιών μας. Και βεβαίως ε, η μειωμένη απορρόφηση. Λόγω του ότι έχουν να κάνουμε 15-20 διαφορετικέ διαδικασίε και νομοθετικές αρμοδιότητες. Ας πούμε στην υγεία είχαμε 500 προγράμματα με κόστος κάτω από 1 εκατομμύριο ευρώ. Και αυτό έναντι 22 διαφορετικών νομοθετικών περιβαλλόντων. Αυτά είχαν να αντιμετωπίσουν οι εταίροι μα οι αποδέκτε τη βοηθεία. Οπότε, δεν θα ήταν χρήσιμο για να παρατρύνουμε τα κρατημέλη να βελτιώσουν την κατανομή της εργασίας να εξειδικευθούν οι χώρες μας ως δωρητές. Γιατί κάποιοι δωρητές έχουν αναπτύξει καλές πρακτικές σε κάποιους τομείς. Θα ήταν λοιπόν σκόπιμο πιστεύω να τους επιτρέψουμε αυτοί να κινηθούν πιο δραστήρια στο συγκεκριμένο τομέα στο πλαίσιο μιας ολοκληρωμένη πολιτικής και με γνώμονα την καταλύτερη κατανομή τη εργασία. Μήπω λοιπόν να ενθαρρύνουμε την εξειδίκευση ή εν πάση περιπτώσει την αξιοποίηση των καλών πρακτικών στον ένα ή τον άλλο τομέα από συγκεκριμένου δωρητέ. Δεύτερον, πριν από μερικά χρόνια στην Κομισιόν είχε δημιουργηθεί ένα άτλα δωρητών, χορηγών βοήθεια. Όπου ο καθένα είχε καταγράψει τι ανάγκε του, τι δυνατότητέ του, αυτός ο άτλας, ο χάρτης αν θέλετε, επέτρεπε στον Επίτροπο να έχει μια γενική εικόνα του ποιος κάνει τι για να αποφύγουμε τις ε, επικαλύψεις και να δούμε ενδεχομένως που υπήρχαν και κενά για να αξιοποιήσουμε καλύτερα την βοήθεια. Ε, κύριε Επίτροπε, όταν ήμουν και εγώ Επίτροπο, θυμάμαι ότι μία από τι δυσκολίε ήταν να έχουμε σε πραγματικό χρόνο τα στοιχεία από συγκεκριμένα κράτη-μέλη τα οποία ήταν αρκετά μυστικοπαθή για κάποιο λόγο όσον αφορά τα επικείμενα σχέδια. Αυτό ο χάρτη ε, χορηγών βοήθεια εν πάση περιπτώσει, πρέπει να παραμείνει λειτουργικό. Τρίτον, θα πρέπει να συνεργαστούμε όχι μόνο μεταξύ μα ή με την Κομισιόν, αλλά και με τρίτου χορηγού βοήθεια, τρίτε χώρε. Έχω στο μυαλό μου άλλου, α πούμε, για παράδειγμα, διεθνεί οργανισμού γιατί όχι. Και τέταρτον, οι πόροι. Θεωρώ, θα το πω, ότι ορισμένα κράτη-μέλη συμπεριφέρονται με σκανδαλώδη τρόπο. Το 2005 τα κράτη-μέλη μας δεσμεύθηκαν για το 0,5% το 2010. Ήταν σε ενδιάμεσος και μόνο στόχος για να μπορέσουμε να προχωρήσουμε και να πάμε ψηλότερα. Και είμαστε στο μισό αυτού του στόχου. Τίποτα δεν πετύχαμε λοιπόν. Είμαστε στο 0,39. Από το 2010, επαναλαμβάνω, έπρεπε να είμαστε στο 0,56. Και κάτι άλλο το οποίο με ανησυχεί γιατί μιλάμε πολύ για τον φόρο επί των χρηματοπιστωτικών συλλαγών. Όμως και εκεί χάσαμε το αντικείμενο με τρόπο σκανδαλώδη. Όταν ακούστηκε για πρώτη φορά αυτή η ιδέα, ο στόχος του μέτρου ήταν να χρησιμοποιήσουμε τους πόρους για την ανάπτυξη, να βοηθήσουμε τις αναπτυσμένες χώρες. Αυτό έχει ξεχαστεί στις μέρες μας. Πού θα πάνε αυτά τα έσοδα. Θα βοηθήσουν τους εθνικούς προπολογισμούς. Και δεν θα με ακρηγορήσω, διότι η κυρία Πρόεδρος είναι αυστηρή και καλός. Αυτά είναι όμως τα στοιχεία που θέλω να καταθέσω καταρχήν. Ευχαριστώ πολύ, Λίλη Πρόεδρος. Όντως ο χρόνος ε, είναι πολύ περιορισμένος. Παρακαλώ να είστε όλοι σύντομοι σε δύο λεπτά. Κύριε Λόρα Γιόγκ, παρακαλώ. Thank you very much, Chair. Κύριε Πρόεδρε, να πω καταρχήν ότι συμφωνώ με τον Επίτροπο. Είμαι από την Βουλή των Λόρδων, από το Ηνωμένο Βασίλειο. Χάρηκα που τον άκουσα να λέει ότι η ειρήνη και η εφορία δεν είναι δυνατές χωρίς την βοήθεια. Χρειάζεται διαφάνεια στο εμπόριο και όχι αποφύγη της φορολογίας. Οι συνθήκες βεβαίως έχουν αλλάξει σε σχέση με το παρελθόν. Ας προσέξουμε λοιπόν πώς χρησιμοποιούμε τις λέξεις. Δεν μιλάμε για δωρητές, για χορηγούς βοήθειες αν θέλετε και αποδέκτες, αλλά δεν νομίζω ότι αυτό βοηθάει το θέμα. Για να το σκεφτούμε και αυτό, τη γλώσσα που χρησιμοποιούμε λοιπόν, ε, θα ήθελα να αλλάξουμε τη δική μας αντίληψη για να αλλάξει και η αντίληψη του κοινού για το θέμα. Μετά θα μπορούσε να μας πει ο Επίτροπος για το ρόλο των ΜΚΟ και της κοινωνίας των πολιτών στην ανάπτυξη και ιδιαίτερα των φορέων που έχουν την έδρα τους στις λεγόμενες χώρες αποδέκτες της βοήθειας. Πρόεδρος, ευχαριστώ πολύ. Και ζητάνα, ε, Βέλγιο, παρακαλώ. François de Donéa, je sais que c'est difficile à prononcer, mais on sait que François de Donéa πρόεδρος της Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων της Βουλής των Αντιπροσώπων του Βελγίου κύριε Πρόεδρε. Συγχαρητήρια καταρχήν για την σημερινή συνάντηση. Σύμφωνα απολύτω με τον Επίτροπο, το μόνο που θα πω λοιπόν είναι τα δύο εξή. Γιατί ούτω ή άλλω θα έρθουμε αργότερα στο δεύτερο θέμα. Πρώτον, όσον αφορά την συνοχή των πολιτικών βοήθειας και την διαφάνεια, τα είπε βεβαίω ο Επίτροπο, μίλησε για την εκμετάλλευση των δασών κλπ. Έχει μεγάλη σημασία η Ευρωπαϊκή Ένωση να αγωνιστεί πιο αποτελεσματικά κατά της ε, στοχευμένης διαφθοράς εκ μέρους των ευρωπαϊκών εταιριών που εκμεταλλεύονται φυσικούς πόρους. Έχουμε εισηγμένες εταιρείες, ευρωπαϊκές εταιρείες, οι οποίες λαδώνουν στις χώρες, σε αναπτυσσόμενες χώρες για να πετύχουν τους στόχους τους. Πρέπει επίσης να ενθαρρύνουμε τον ΩΣΑ να εντείνει τι προσπαθίε του προς την διακατεύθυνση και με τις χώρες BRIC να κάνει ό,τι μπορεί ώστε να καταπολεμηθεί η διαφθορά. Γιατί αυτό είναι η μεγάλη αντίφαση στην πολιτική μας. Η διαφθορά είναι το ένα πράγμα και μετά πέρα από την συνοχή έχουμε και το θέμα της αποτελεσματικότητας. Πολύ σημαντικό. Έναντι των φορολογουμένων μας, οι οποίοι έχουν βαρεθεί, για να μην πω ότι δεν έχουν καμία όρεξη πλέον να πληρώνουν, όταν βλέπουν ότι Κάποιοι δωροδοκούν στις αναπτυσσόμενες χώρες για να πετύχουν τους στόχους τους. Τώρα όσον αφορά τα τοπικά κοινοβούλια και την ενημέρωσή τους, πώς ενημερώνονται για την βοήθεια που τους δίνουμε. Ο Ρουι Μισελ αναφέρθηκε στην Τανζανία, με εκατοντάδες έργα, ο Πίτροπος είπε για το Μαλάουι, αν δεν κάνω λάθος. Όταν συναντώ βουλευτές τρίτων χωρών, παραπονούνται για το ότι οι κυβερνήσεις δεν τους ενημερώνουν για τα ποσά τα οποία λαμβάνουν και τα οποία δεν εμφανίζονται καμιά φορά στον προπολογισμό. Πρέπει λοιπόν στις χώρε αυτές να βελτιώσουμε την διαφάνεια και τη συνοχή εννοείται και να φροντίσουμε κάθε φορά που υπογράφουμε μια σύμβαση χωρίς βοήθεια Πρόεδρος, ε, με συγχωρείτε, είπα δύο λεπτά ε, κύριε Τεντονεά ενισχύσουμε λοιπόν τον ρόλο των Εθνικών Κοινοβουλίων στις χώρες αποδέκτες της βοήθειας. Αυτό είπε ο κ. Δονεά. Ευχαριστώ Πρόεδρε και εγώ Λέω ο κύριος Κορτές Λάστρα. Και εγώ θέλω να σας ευχαριστήσω για την ε, διοργάνωση αυτής της συνεδρίασης. Ε, Παρ' το λόγο για να ε, πω ότι συμφωνώ απόλυτα με τον κύριο Πιμπάλξ τα πολλαπλά ταξίδια προς διάφορους τόπους όπου αναπτύσσονται τα σχέδια αναπτυξιακής συνεργασίας μπορούσαμε να δούμε αυτό το κοινοπρογραμματισμό, πώς εξελίχθηκε και πώς υπάρχει ήδη μια σαφής ιδέα ότι πρέπει να υπάρχει ένας κοινό προγραμματισμός για να έχουμε καλύτερα αποτελέσματα για το σύνολο των χωρών. Όμως εξακολουθούμε να έχουμε πολλές επιφυλάξεις από αρκετά κράτη-μέλη για να γίνει κάτι τέτοιο. Εγώ ελπίζω ότι με τη δική σας προσπάθεια και την προσπάθεια όλων θα το πετύχουμε σιγά σιγά. Θα ήθελα να κάνω και μια σκέψη για ένα άλλο θέμα. Εσείς ε, αναφερθήκατε στο ότι η αναπτυξιακή βοήθεια δεν είναι στο παγιό της αυτή τη στιγμή, ακριβώς γιατί κάποια κράτη-μέλη δεν έχουν τηρήσει τις δεσμεύσεις τους ε, αλλά εγώ θα ήθελα να εσείς να τονίσετε ιδιαίτερα αυτό το διπλό φαινόμενο. Δηλαδή, κάποιες ε, χώρες ε, ε, ουσιαστικά μειώνουν την αναπτυξική βοήθεια με για κατόπιν έρχονται στις Βρυξέλλες και ζητούν να έχουμε ισχυρή αναπτυξική βοήθεια. Ας είμαστε λοιπόν ε, συναφείς και απέναντι στη στάση που έχουμε σε, σε αυτά τα κράτη-μέλη. Έτσι λοιπόν, θέλω να κάνω μια ερώτηση και ένα αίτημα ξεκινώ με το θέμα της ε, πολιτικής συνοχής και της συνεργασίας Βορρά-Νότου. Θα ήθελα να συζητήσω σε αυτές τις ε, στιγμές ε, που βιώνει η συνεργασία και εσείς ε, ως Επιτρόπος θα το ξέρετε αυτό, κάποιος θα μπορούσε να σκεφτεί να ελαχιστοποιήσει, να υποβαθμίσει την ε, έννοια ε, της συνεργασίας, γιατί εμείς οι βουλευτές έχουμε την αντίθετη υποχρέωση, όπως είπε και ο κύριος Μέτσιλ, δηλαδή να ενισχύσουμε την συνεργασία σε αυτές τις στιγμές, δηλαδή πέρα από την κρίση που βιώνουμε αυτούς τους καιρούς. Μάλιστα, σας ευχαριστώ. Ο κύριος Άντζελ από το Λουξεμβούργο. Για μισή λεπτό. Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τον Επίτροπο για τη δεσμευσή του εντός των Ηνωμένων Εθνών και για την ομάδα που θα προετοιμάσει τους αναπτυξιακούς στόχους της χιλιετίας για μετά το 2015 και επίσης να συγχωνευτούν αυτοί οι στόχοι με τους στόχους της αηφόρου ανάπτυξης. Είχαμε, είδαμε μια ενδιαφέρουσα ανακοίνωση πριν ένα μισή μήνα από την Κομισιόν και εγώ νομίζω ότι αυτό είναι ένα πάρα πολύ μεγάλο βήμα προς τη συνοχή των πολιτικών. Να ρωτήσω, σε αυτή τη διαδικασία έχει σημειωθεί κάποια πρόοδος. Εσείς πιστεύετε ότι οι ιδέες που μας παρουσιάσατε στην ανακοίνωσή σας εντός των Ηνωμένων Εθνών ε, θα βρουν κάποια διέξοδο, θα σημειωθεί κάποια επιτυχία, γιατί όπως σας είπα έχουμε ένα πολύ μεγάλο βήμα προς τη συνοχή εδώ και θα ενημερώσω τον Επίτροπο ότι χτε ε, στην συνεδρία τη Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων αποφασίσαμε να σα καλέσουμε στην Επιτροπή μα για να συζητήσουμε για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Ανάπτυξη. Δυστυχώ ε, πάντοτε βρίσκεται εκτό του Ευρωπαϊκού Προπολογισμού και σκεφτήκαμε λοιπόν ότι θα ήταν ενδιαφέρον να συζητήσουμε μαζί σας για το Ταμείο αυτό για να έχουμε μια καλύτερη εικόνα και για να μπορέσουμε να κάνουμε και ένα μικρό κοινοβουλευτικό έλεγχο επί αυτού του πολύ σημαντικού ταμείου. Σας ευχαριστώ για το λόγο, Πρόεδρε. Πρόεδρος, θα δώσω τώρα το λόγο στην κυρία Μπάιερ από την Αυστρία. Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε. Λέγομαι Μπάιερ. Είμαι πρόεδρος της Επιτροπής για την Ανάπτυξη στο Αυστριακό Κοινοβούλιο. Υπάρχει μια οδηγία πρόσφατη αν θέλετε της Ευρωπαϊκής Επιτροπής που αναφέρεται στην ε, εταιρική κοινωνική υπευθυνότητα ε, και η οποία ε, αφορά δεν αναφέρεται αν θέλετε στη, σε αυτά τα κριτήρια τα οποία θα θέλαμε να υπάρχουν εδώ για την ανάπτυξη. Θα έπρεπε να υπάρχουν και εδώ κριτήρια και να αναλαμβάνουν δεσμεύσει οι εταιρείε. Οι ευρωπαϊκές εταιρείες ξέρουμε ότι εφαρμόζουν πολιτικές οι οποίες, τις οποίες δεν θα ε, υποστηρίζαμε οι οποίες ε, δεν είναι διαφανείς ε, λάβετε υπόψη σας επίσης ότι ιδιαίτερα για τα βιοκαύσιμα και τα λοιπά για την αρπαγή στην Αφρική και όλα αυτά εκεί εμπλέκονται ευρωπαϊκοί ευρωπαϊκές εταιρείες οι οποίες χρησιμοποιούν και χρήματα ταμείων συνταξιδοτικών των Ευρωπαίων πολιτών και δεν δρούν με τον σωστό τρόπο. Κύριε Επίτροπε, ευχαριστώ πολύ για τις παρεμβάσεις σας. Χάρηκα ιδιαίτερα για αυτά που είπατε και εκτιμώ ιδιαίτερα τη δουλειά που κάνετε και αυτή του Μισελ Μπαρνιέ. Να ρωτήσω το εξή τι γίνεται με τους φυσικούς πόρους των αναπτυσσομένων χωρών. Είμαι μόνιμη συγκήτρια για την ανθρωπιστική βοήθεια και βλέπω ότι στις χώρες που έχουν πολλούς φυσικούς πόρους δεν, ε, οι πολίτες είναι φτωχοί δεν ε, αξιοποιούνται προς όφελος των πολιτών αυτοί οι φυσικοί πόροι σε μια συνάντηση με τις χώρες ΑΚΕ ήταν και ο Λουί Μισελ παρόν συζητήσαμε το θέμα αυτό εσείς τι νομίζετε και τι θα γίνει με το μέλλον της Συμφωνίας Κοτονού Τελευταίος ομιλητής, ο κύριος Πίσκο, Πορτογαλία. You have the floor. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Θέλω να θέσω δύο ερωτήσεις. Καταρχήν, ποιο είναι το επίπεδο συνεργασίας μεταξύ των κρατών μελών και μεταξύ τους αλλά και με την Ευρωπαϊκή Ένωση σε ό,τι αφορά στο συντονισμό των ε, αναπτυξιακών πολιτικών και κυρίως ε, βλέποντας την τάση ότι πάρα πολλές χώρες έχουν πολύ συγκεκριμένα συμφέροντα σε πλαίσια μιας διμερούς συνεργασίας ε, με χώρες που αναπτύσσουν project. Δεύτερη ερώτηση. Σε ποιο βαθμό υπάρχει συνεργασία με τρίτες χώρες όπως με την Κίνα ή τη Βραζιλία που είναι σημαντική εταιρεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Βλέπουμε αυτή τη συνεργασία λοιπόν γιατί ξέρουμε ότι υπάρχουν ε, ουσιαστικά κάποιες απώλειες. Ε, έτσι λοιπόν θα ήταν σημαντικό να δούμε αν μπορούμε να έχουμε ένα επίπεδο διαλόγου με τις χώρες αυτές. Σας ευχαριστώ. θα σας δώσω το λόγο κύριε Πίμπαλξ για να απαντήσετε όλες αυτές τις ενδιαφέρουσες ερωτήσεις. Θα προσπαθήσω να είμαι σύντομος για την εξειδίκευση αν θέλετε των χορηγών βοήθειας. Συμφωνώ ότι υπάρχουν οργανισμοί ανάπτυξης όπως και η ΤΕΖΕΤ παραδείγματος χάρη και άλλες και άλλοι οργανισμοί που υπάρχουν και που έχουν κάποια αν θέλετε ειδικότητα σε ορισμένα πράγματα ε, δεν ξέρω κατά πόσον είναι σωστό να πούμε ότι η Γερμανία ας πούμε θα ασχολείται με την υγεία και μια άλλη χώρα με τη γεωργία δεν είμαι σίγουρος ότι είναι καλό να το κάνουμε αυτό έτσι και αλλιώς για πολλούς από αυτούς τους ε, οργανισμούς είναι κρατικοί οργανισμοί καλά κάνουν και εξειδικεύονται και βεβαίως θα τους χρησιμοποιήσουμε αλλά σε πολιτικό επίπεδο νομίζω ότι δεν είναι σωστό να εξειδικεύουμε τα πράγματα. Θα πρέπει να έχουμε μια ευρεία προσέγγιση γιατί όλες οι χώρες μπορούν να κάνουν πολλά πράγματα. Τώρα, And ε, βεβαίως έχουμε πολλά προβλήματα ε, βεβαίως με την αναπτυξιακή βοήθεια είναι τα πράγματα χειρότερα από ό,τι στη δική σας εποχή κύριε Μισελ και σίγουρα υπάρχουν προβλήματα συντονισμού και στην Ευρωπαϊκή Ένωση και και στις χώρες προσπαθούμε να βοηθήσουμε. Δεν είναι μοναχά πολιτικό, πολιτικά τα προβλήματα, είναι συστημικά. Τώρα, για την εξωτερική συνεργασία, νομίζω ότι εδώ υπήρξε βελτίωση με οργανισμούς όπως Παγκόσμια Τράπεζα, το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, ιδιαίτερα αυτό το, ιδιαίτερα το Δουνουτού, συνεργαζόμαστε για πολύ ε, συγκεκριμένα θέματα με την Παγκόσμια Τράπεζα τα πράγματα είναι σε πιο πολιτικό επίπεδο με το USAID έχουμε, συνεργαζόμαστε για την διατροφή με την Ιαπωνία ε, για κάποιες χώρες του Ειρηνικού και με τη Γαλλία για τον Νότιο Σουδάν και τα λοιπά. Ε, ε, έχουμε κάνει πρόοδους. Ινδία, Κίνα, Μπραζίλ, είπαμε τις χώρες Μπρίκα, υπάρχουν πολλά κενά ακόμη. Τώρα για το φόρο χρηματοπιστωτικών συναλλαγών. Όντως έχουμε χάσει το τρένο εδώ και συνεχίζουμε να έχουμε χάσει, να χάνουμε ευκαιρίες συνεχώς υπάρχουν προβλήματα εδώ και αυτό σχετίζεται και με τις σχέσεις μεταξύ χορηγών και αποδεκτών είναι, δημιουργούνται προβλήματα και παγίδες και πέφτουμε σε παγίδες εδώ νομίζω ότι εδώ χάνουμε ευκαιρίες όχι επειδή μ' αρέσει ιδιαίτερα ο φόρος χρηματοπιστωτικών συναλλαγών αλλά γιατί δεν κάνουμε, ε, δεν παίρνουμε μέτρα για να ε, μπορούμε να κάνουμε κινήσεις σε παγκόσμιο επίπεδο και όχι με μονομένα με ορισμένες χώρες. Τώρα για τους μη κυβερνητικού οργανισμούς και την κοινωνία των πολιτών ε, συνεχίζουμε να έχουμε ε, σχέσεις και θα συνεχίσουμε εφόσον το επιτρέπουν οι πόροι μας και με τις, την τοπική αυτοδιοίκηση και με και ιδιαίτερα με την κοινωνία των πολιτών γιατί πιστεύουμε ότι ε, σε ορισμένες χώρες ε, ήδη λειτουργούν οι ε, μη κυβερνητικοί οργανισμοί και η κοινωνία των πολιτών ε, και έχουν πολύ καλή συνεργασία. Θα πρέπει να την ενισχύσουμε. Από εκεί και πέρα για την διαφάνεια με τη, στη βοήθεια τα πολλά από τα προβλήματα των, της διαφάνειας προέρχονται από μας. Θα πρέπει οι ροές βοήθειας είναι σαφείς και θα πρέπει να επιμείνουμε στο να είναι σαφείς και ακριβείς. Για του χρόνου ας πούμε το Μαλάουι θα πρέπει να βάλει τη βοήθεια στον προϋπολογισμό του 2014. Αλλά Συνήθω δεν μπαίνει η βοήθεια αυτή καθεαυτή μπαίνει ένα προς υπόμνηση ή ένα ή, και Παραδείγματο χάρη στο Μπουρούντι είδαμε ε, να γίνεται αυτό και να χρησιμοποιούνται οι πόροι για άλλους σκοπούς. Ε, ε, Πρέπει λοιπόν να επιμείνουμε σε αυτό για να είναι διαφανείς οι ροές βοήθειες ε, όπου δεν είναι μόνο μονόδρομος ε, βεβαίως φταίμε κι εμείς πάρα πολύ τώρα για τη συνεργασία βορρά-νότου δεν ξέρω αν πρόκειται για συνεργασία ε, βεβαίως υπάρχουν επενδύσεις που πρέπει να γίνουν σε επτυσσόμενες χώρες για να προχωρήσουν οι χώρες αυτές υπάρχουν όμως και άλλες ε, επενδύσεις εντός εισαγωγικών ε, για χώρες ε, οι οποίες έχουν χαμηλό εθνικό προϊόν αν θέλετε και το οποίο πάνε σε ανεπτυγμένες χώρες και ζητούν βοήθεια δεν είναι σωστό όμως να μιλάμε για συνεργασία βορρά-νότου. Μιλάμε για παγκόσμια συνεργασία. Δεν είναι σωστό να ε, δίνουμε αν θέλετε γεωγραφικούς προδιορισμούς στη βοήθεια τριγωνική υπάρχουν και οι όροι τριγωνική συνεργασία. Ας πούμε, Ο Αυστραλία, Φίτζι, αποδέκτηση είναι το Φίτζι και Ευρωπαϊκή Ένωση είναι τριγωνική συνεργασία υπάρχει τριγωνική συνεργασία αλλά νο, πιστεύουμε ο, πιστεύω ότι αυτή η ιδεολογική προσέγγιση σαν να υπάρχει υπάρχει διαφορά μεταξύ αν θέλετε ορισμένων κάποια συνεργασίας βορρά νότου, νότου, νότου και τα λοιπά ε, δεν είναι σωστό η, η, συνεργασία και βοήθεια είναι η ίδια παγκοσμίω από όπου και αν προέρχεται προς όποιον και να πηγαίνει τώρα για τα εθνικά κοινοβούλια και για την, α, τις προσκλήσεις να πάω σε εθνικά κοινοβούλια εξαρτάται βέβαια και από το πρόγραμμα πρόγραμμά μου βεβαίως αλλά δεν έχω καμία αντίρρηση να τα, επισκεφθώ τα εθνικά κοινοβούλια τώρα για τους φυσικούς πόρους ε, και τη φτώχεια και εδώ σημαντικό είναι η διαφάνεια. Όλα ξεκινάνε από τη στιγμή που ε, φτιάχνεται η σύμβαση. Μόνο μετά από αυτό πάνε τα χρήματα στις κυβερνήσεις και η πρώτη απέτησή μας είναι η διαφάνεια. Όταν έρχεται, έρχονται τα χρήματα θα πρέπει να μπουν στο προϋπολογισμό και θα πάνε για αυτό το σκοπό ή ετοιμάζουμε μια σχετική οδηγία η οποία θα περάσει ως το δυνατόν πιο γρήγορα. Τώρα για τη, συν, για τη φορολογική συνεργασία Υπάρχει εδώ ένα συγκεκριμένο κονδύλι από το ΑΕΜΕ για την υποστήριξη των εφοριών και των για τη φορολογική διοίκηση αλλά δεν είδαμε καν δεν υπάρχει αίτημα σχετικά τώρα για το κοτονού με, ε, αυτή τη στιγμή διανύουμε μια περίοδο περισυλλογή. θα δούμε τι θα γίνει το 2020 δεν μπορώ να απαντήσω τίποτα παραπάνω σχετικά για το τι θα γίνει με την Κοτονού από εκεί και πέρα για το επίπεδο συνεργασίας των χωρών μελών νομίζω ότι έχουμε φτάσει στο μάξιμουμ ανταλλαγή πληροφοριών και διαφάνειας με τα κράτη-μέλη. Ε, το επόμενο βήμα είναι ο κοινό προγραμματισμός. Ο τρόπος με τον οποίο δρούμε τώρα ίσως δεν είναι πολύ υπεύθυνο διότι εδώ διαχειριζόμαστε χρήματα του φορολογουμένου έτσι δεν μπορούμε να, σπατά, να διασπαθίζουμε τους πόρους αυτούς είναι τους χάνουμε δεν μπορούμε να αποτύχουμε είναι τα χρήματα των φορολογουμένων αυτό και κάθε ευρώ που επενδύνουμε είτε προέρχεται το ευρώ από τη Λετωνία είτε προέρχεται από τη Γερμανία είτε από οπουδήποτε προέρχεται θα πρέπει το κάθε ευρώ που επενδύεται να στοχεύει στις ανάγκες της συγκεκριμένης χώρας και να μπορεί να αποδώσει καρπούς. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πίμπαλξ, λέει η κυρία Ζολή, ε, που μας παρουσιάσετε τη θέση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Καθίσατε και λίγο παραπάνω από ό,τι προβλεπόταν. Θα δώσω τώρα το λόγο στον κύριο Γκέρ, την Προεδρία, στον κύριο Γκέρενς, γιατί θα προεδρεύσει αυτό το τμήμα της συνάντησης. Euh, Ευχαριστώ, Εύα Ο χρόνος ε, πιέζει πάρα πολύ. Υποτίθεται ότι θα ξεκινήσουμε 9.45 για να τελειώσουμε 10.55. Ξεπεράσαμε τον χρόνο για την πρώτη συζήτηση κατά 30 λεπτά. Οπότε αντιπαρέχομαι τα εισαγωγικά σχόλια και περνώ κατευθείαν στην ανταλλαγή απόψεων με τα Εθνικά Κοινοβούλια. Κοιτάξτε, ήρθαμε εδώ για να ακούσουμε εσά. Οπότε, επαναλαμβάνω ότι δεν θα προβώ σε εισαγωγή. Ε, να ξεκινήσουμε με τον κύριο Westcott, το οποίο ε, εκπροσωπεί την υπηρεσία εξωτερική δράση και μετά έχουμε Ισπανία, Ουγγαρία, Πορτογαλία, Ηνωμένο Βασίλειο. Παρακαλώ, πέντε λεπτά ο καθένα ε, αυτό ήταν το αρχικό βεβαίω. Θα έλεγα τέσσερα λεπτά και, και εσείς κύριε Westcott παρακαλώ να είστε εξαιρετικά σύντομος για να μην απογοητεύσουμε και τους εκπροσώπου των Εθνικών Κοινοβουλίων. Ε, μια λέξη μόνο όσον αφορά τον ορισμό της συνοχής των πολιτικών. Συνοχή σημαίνει να μην ε, κατεδαφίζει ο ένας αυτό το οποίο οικοδομεί ο άλλος. Αν το καταφέρουμε αυτό, ήδη θα προλάβουμε λάθη σε πολλούς τομείς. Κύριε Westcott, παρακαλώ. Πείτε μας πώς βλέπει το θέμα η υπηρεσία εξωτερικής δράσης. Πρόεδρε, αντιλαμβάνομαι ότι ο Επίτροπος έπρεπε να φύγει γιατί είχε άλλη συνεδρίαση. Εγώ θα είμαι σχετικά σύντομο, διότι τα περισσότερα ζητήματα που συζητούμε τα καλύψαμε τόσο επίτροπο ο και μάλλον συμφωνούμε. Οπότε, τώρα, η... ο ρόλος μας στην ανάπτυξη απορρέει από τις οδηγίες που έχουμε λάβει από τα κράτη-μέλη που μας είπαν ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να εξασφαλίζει συνοχή μεταξύ τη ανάγκη εξωτερική εξωτερικής βοήθειας και των άλλων πολιτικών. Η εξωτερική δράση, με άλλα λόγια, πρέπει να λαμβάνει υπόψη τη την πτυχή ανάπτυξη. Ο ρόλο τη υπηρεσία μα είναι ένα και ενιαίο και περιέχει ακριβώ την προσπάθεια να βοηθήσει την ανάπτυξη ανά τον κόσμο. Εγώ εξειδικεύομαι στην Αφρική και θα σας δώσω συγκεκριμένα μερικά παραδείγματα του πώς συγκεκριμένα υλοποιούμε τη δράση μας στην Αφρική. Η συνοχή των πολιτικών είναι ενταγμένη στο DNA μας, θα έλεγα, της υπηρεσίας μας. Όχι μόνο για τους σκοπούς της ανάπτυξης, αλλά και εν γέννη, θα έλεγα, σε όλες τις πολιτικές μας, ε, εμπόριο, περιβάλλον, κοινωνική πολιτική κλπ. Σε όλες τις δραστηριότητες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Από την εμπειρία μου στην Αφρική και στην Ευρώπη και σε άλλες χώρες, πρέπει να σας πω ότι η σχέση ασφάλεια και ανάπτυξη είναι κρίσιμη σημασία. πρέπει να τη λάβουμε υπόψη μα αν θέλουμε να πετύχουμε του στόχου μα. Η συνοχή αυτή, η αυτοσυνέπεια αν θέλετε, εκφράζεται με πολλού τρόπου. Πρέπει να υπάρχει καταρχήν αυτοσυνέπεια μεταξύ αυτών που κάνουμε εμεί και τα διάφορα θεσμικά όργανα, η Επιτροπή, η Επίτροπη, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Εσωτερική λοιπόν συνέπεια, αν θέλετε. Και πρέπει να υπάρχει και συνοχή και συνέπεια με τις πολιτικέ των κρατών μελών. Έτσι όπω υλοποιούνται αυτέ σε διάφορε φορές τη Αφρική. Αλλά υπάρχει και συμβατότητα με τι δράσει άλλων φορέων. Είχαμε πάει και είχαμε δει την περσμένη εβδομάδα το ΔΕΛΤΑΝΙΤΑΦ, την Παγκόσμια Τράπεζα και είπαμε κάτι να κάνουμε συλλογικά και συντονισμένα. Τρίτον, εξίσου σημαντικό, αυτό συνέπεια ε, και συνέπεια στη σχέση μας με τους Αφρικανούς εταίρους. Διότι Η σχέση, όπω είπαν και άλλοι, πρόκειται για εταιρική σχέση, όχι για απλή χορήγηση βοήθεια σε αποδέκτε, λήπτες. Έχουμε λοιπόν την Αφρική Ένωση, την ECOWAS, την SADEC, έχουμε και άλλου συλλογικού φορεί, αλλά και τι χώρε τις ίδιες. Και στι χώρε, βέβαια, μην ξεχνάτε ότι δεν μιλάμε μόνο με την κυβέρνηση, αλλά με την κοινωνία των πολιτών, με τι επιχειρήσει, γιατί χωρί και την δική του συμμετοχή και πάλι δεν θα πετύχουμε του στόχου μα. Όλα αυτά συμπληρώνονται σε αυτό το οποίο λέει και είπατε εκπρόσωπος ε, χρειαζόμαστε μια αυτοσυνεπή προσέγγιση για να αντιμετωπίσουμε να καλύψουμε τις ανάγκες αυτών των χωρών και θα σας δώσω τρία παραδείγματα από την Σομαλία το Σαχέλ και το Σουδάν Σομαλία κλασικό παράδειγμα όπου πριν την υπηρεσία μας η Ευρωπαϊκή Ένωση παρενέβαινε με τρόπο αποσπασματικό στη Σομαλία, στο Βορρά, κυρίως είχαμε ένα πολύ σημαντικό πρόγραμμα. Είχαμε και την ανθρωπιστική παρέμβασή μας, είχαμε παρουσία στρατιωτική για να αντιμετωπίσουμε τα φαινόμενα πειρατείας με την ενίσχυση της ε, Αφρικανικής Ένωσης. Είχαμε και μια παρουσία για την εκπαίδευση των δυνάμεων της κυβέρνησης της Σομαλίας. Αλλά όλα αυτά αποσπασματικά, επαναλαμβάνω υπηρεσία εξωτερικής δράσης, τα μάζεψε όλα αυτά, τα συντόνισε και τα ενέταξε σε μια ευρύτερη στρατηγική για το κέντρο της Αφρικής. Για να πετύχουμε όλοι μαζί συγκεκριμένους πια στόχους. Συνεργαζόμαστε πλέον με τη νέα μόσπονδη κυβέρνηση της για να τα, θέσουμε, να κάνουμε αυτά πράξη και υπάρχει πλέον και ένα σύμφωνα αν θέλετε μεταξύ τη νέα κυβέρνηση και τη διεθνού κοινότητα. Όλοι μαζί κάνουμε ό,τι μπορούμε, ό,τι καλύτερο μπορούμε για να υποστηρίξουμε τη Σομαλία να πετύχει ανάπτυξη και ασφάλεια στη χώρα. Στο Σαχέλ και προκειμένου στο Μάλι. Και εκεί είδαμε ακριβώ το ίδιο πρόβλημα. Μπορούμε να βοηθήσουμε φυσικά το Μάλι. Τα κεφάλαια τα τελευταία δέκα χρόνια προς το Μάλι ήταν πολύ μεγάλα για την εκπαίδευση, το περιβάλλον, την κοινωνία, την οικονομία. Και όμω. Όλα αυτά μπορούν να πανεστράφει αν δεν έχουμε την κατάλληλη πολιτική κατάσταση και, και ασφάλεια. Τα παιδιά δεν μπορούν να πάνε σχολείο αν δεν υπάρχει ασφάλεια. Ε, αν ε, δίνουμε λεφτά για νοσοκομεία και κλινικέ και λελατούνται, ε, στο τέλο δεν πετυχαίνουμε τίποτα. Μπορούμε λοιπόν με την ανάπτυξη να πετύχουμε πολλά, και μεταξύ άλλων και ασφάλεια, αλλά ισχύει και το αντίστροφο χωρί ασφάλεια. Δεν μπορούμε να βελτιώσουμε τι συνθήκε ζωή των ανθρώπων στην περιοχή. Αλλιώς οι άνθρωποι θα εμπλακούνται σε πολεμικέ δραστηριότητε, λατρεμπόριο και οτιδήποτε άλλο. Και όλα αυτά, και για άλλη μια φορά, παραλαμβάνω ότι έγιναν κομμάτι μια ευρύτερη στρατηγική. Εμείς στο Μάλι συγκεκριμένα δεν καταφέρουμε να εξασφαλίσουμε τη συνεργασία των εταίρων της περιοχής. Προσπαθούμε όμως και σήμερα, όχι μόνο με γνώμονα την ανάπτυξη στην περιοχή αλλά και στις γειτονικέ χώρες, αλλά και με γνώμονα την ασφάλεια. Έχουμε την EU Camp Sahel, ε, βοηθούμε τον Νίγηρα να μην αντιμετωπίσει τα προβλήματα που αντιμετωπίσει το Μάλι, το ίδιο στην Μπουρκίνα Φάσο και στην Μαυρτανία. Η συνεργασία λοιπόν μεταξύ του Επιτρόπου και της υπηρεσία μας είναι πολύ στενή. Επίσης το EDF χρηματοδοτεί το χρηματοδοτικό εργαλείο για την Αφρική και θα δώσουμε έτσι τη δυνατότητα στους Αφρικανούς να πάρουν στα χέρια τους την ασφάλειά τους. Στη Σομαλία έχουμε την Amazon και τώρα την Έχουμε τη δύναμη αφίσμα, όπως λέγεται, τη δύναμη στο Μάλι που υποστηρίζει τις γαλλικές στρατιωτικές δυνάμεις. Στο Σουδάν, εκεί που γεννήθηκε η ολοκληρωμένη προσέγγιση μας, στο νέο Σουδάν, έχουμε μια νέα χώρα, μια τελείως νέα χώρα. Μια χώρα η οποία οικοδομείται εκ του μηδενό. Και εκεί καταρτήσαμε μια πολιτική ολοκληρωμένη, η οποία ενσωματώνει όλα τα επιμέρους στοιχεία της παρέμβασης της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και αυτό σε συνεργασία με τα κράτη-μέλη. Εδώ όλοι αυτοσχεδιάζουμε εκ του μηδενός, αλλά πρέπει να αποδείξουμε ότι η συλλογική δράση θα ωφελήσει περισσότερο από οτιδήποτε άλλο το λαό του Σουδάν. Η κατάσταση φυσικά στην περιοχή είναι δραματική, οι ανάγκε είναι τεράστιε και γι' αυτό κάνουμε ό,τι μπορούμε για να υποστηρίξουμε την Αφρικανική Ένωση να επιλύσει τα εκκρεμή ζητήματα μεταξύ Βορρά και Νότου. Πρόκειται μια αντιπαλότητα, με σύραξη που έχει να σοβεί στην περιοχή, στον, ε, στην περιοχή του Γαλάζιου στον Άνω Αυτά τα τρία παραδείγματα τα ανέφερα για να σας τονίσω πόσο στενά συνδεμένα είναι θέματα όπως η ασφάλεια αλλά και το περιβάλλον. Από το Σαχέλ από τη, μέχρι τη Σομαλία και από τη Σομαλία μέχρι την Δυτική Σαχάρα. Όλα αυτά επηρεάζονται μεταξύ άλλων από την αλλαγή του κλίματος. Και αυτό το λαμβάνουμε υπόψη μας ως ε, υπηρεσία εξωτερικής βοήθειας στην προσπάθεια μας να συμβάλλουμε στις ε, διαπραγματεύσεις και στις επιτόπου δράσεις για να αλλάξουμε την πραγματικότητα. Και υπάρχουν πολλά τέτοια παραδείγματα. Η υπηρεσία μας και το πνευματικό σας ετοιμάτων συμβάλλει στον προγραμματισμό για τους σκοπούς της συνοχής και της συνέπειας, όπως είπα. Και συνεργαζόμαστε με τον Επίτροπο στενά αυτή τη στιγμή ακριβώς για να καταρτήσουμε ένα πρόγραμμα τόσο εθνικό όσο και σε περιφερειακό επίπεδο, στο πλαίσιο του EDF που ανέκριναν τα κράτη-μέλη. Και αν θέλετε θα απαντήσω ερωτήσει από αυτού αργότερα. Επίσης, καθώς πλησιάζουμε στο τέλος των διαπραγματεύσεων για τις ε, συμφωνίες εταιρική σύμπραξη, εδώ ο Επίτροπος θα μας βοηθήσει να κλείσουμε αυτέ τι διαπραγματεύσει. Άρα λοιπόν, το ξαναλέω, ε, συνεχίζουμε να είμαστε υπέρ Τη ολοκληρωμένη προσέγγιση και τη συνοχή και τη αυτοσυνέπειας ακριβώ τη δράση μας. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ για τις, ε, τα όσα μας είπατε. Μιλήσατε πολύ για την Δυτική Αφρική και για το Σαχέλ. Και θα δώσουμε το λόγο στον κύριο Ντονέ, ο οποίος εκπροσωπεί και το Βελγικό Κοινοβούλιο. Σας ευχαριστούμε που είστε εδώ μαζί μας και όπως σας είπα θα δώσω το λόγο στους εκπροσώπους τεσσάρων εθνικών κοινοβουλίων, Ισπανία, Ουγγαρία, Πορτογαλία και Ηνωμένου Βασιλείου, για να μας παρουσιάσουν τις απόψεις τους σε σχέση με τη συνοχή των πολιτικών και κατόπιν θα καλέσω τον εκπρόσωπο του Ισπανικού Κοινοβουλίου να είναι πάρα πολύ σύντομος για να μπορέσουμε να δώσουμε το λόγο και στους υπόλοιπους συνάδελφους. Παρακαλώ. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Η Ισπανία έχει συμπεριλήψει στην ομοθεσία της ε, την συνοχή της αναπτυξιακής πολιτικής. Continuez, s'il vous plaît. Συνεχίστε, παρακαλώ. Εγώ δεν άγγιξα τίποτα. Λοιπόν, η συνοχή της αναπτύξική πολιτική ε, στην Ιστάνια έχει συμπεριληφθεί στην νομοθεσία από την ε, έγκριση τη νομοθεσία 93 93-28 και έχουμε μία εντολή που υποχρεώνει όλες τις δημόσιες δικήσεις ε, στο άρθρο 4 αναφέρονται όλες οι αρχές, οι πολιτικές που εφαρμόζουν οι δημόσιες αρχές. No tengo prisa. A pesar Λοιπόν, οι δημόσιες δικήσεις είναι αρμόδιες ε, για την εφαρμογή των διεθνών πολιτικών, όμως ε, όλοι οι δίκες είναι αρμόδια για την, ανάπτυ... για την εφαρμογή της αναπτυξιακής πολιτικής. Άλλες ε, πρωτοβουλίες είναι το σύμφωνο κατά της ανέχειας που έχει υπογραφεί από το Κοινοβούλιο την Κοινωνία των Πολιτών. Además, Πρόσθετα, η Ισπανική Συνεργασία ε, τα τελευταία χρόνια έχει λάβει υπόψη τις ανησυχίες και τις συστάσεις των διεθνών οργανισμών όπως τα Ηνωμένα Έθνη και ο ΟΣΑ και αυτό φαίνεται στη σημερινή θητεία. Ανέφερε ο πρόεδρος Ραχώη στο τελευταίο ομιλία του ε, για την επιστηστική ασφάλεια το θέμα αυτό και εκεί αντικατοπτρίστηκε η στρατηγική μας για τη συνεργασία που θα εφαρμοστεί και σε πάρα πολλούς τομείς όπως το σχάρι το Συμβούλιο Αναπτυξιακής Συνεργασίας y comisiones, el Grupo Και μεταξύ αυτών και η ομάδα εργασία του CDP που δημιουργήθηκε το 2005. Έχουμε επίσης τομείς ε, συντονισμού, τεχνικού συντονισμού υπάρχει και στην ε, γραμματεία της ε, Συνεργασίας για την Ανάπτυξη ένας συντονισμός των πολιτικών τόσο σε διεθνές επίπεδο όσο και σε εγχώριο συνοχή των πολιτικών αποτελεί τμήμα της συνεργασίας που θα σχεδιαστεί για την επόμενη περίοδο που αντικοτοπτρίζεται στην περίοδο 2013-2016. Η Ισπανία είχε σχεδιάσει το τέταρτο σχέδιο προκειμένου να επικεντρωθεί σε μεγαλύτερη συνοχή των πολιτικών. Θέλουμε να ενισχύσουμε τους μηχανισμούς για να βελτιώσουμε τη συνοχή της αναπτυξίας πολιτικής. Ε, το σημερινό σχέδιο προωθεί ε, άμεσες ξένες επενδύσεις και θέτει την ανάγκη να έχουμε επίπτωση στις δράσεις που ακολουθούν οι ισπανικές επιχειρήσεις και επίσης θέλουμε να ενδυναμώσουμε το διάλογο μεταξύ των Υπουργείων υπό την αιγίδα του Υπουργείου Εξωτερικών. Το σχέδιο προτείνει να εργαστούν σύμφωνα με τις κατητηρίες γραμμές της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Θέλουμε μία δημόσια πολιτική διεθνούς ανάπτυξης ε, και γι' αυτό επικεντρώνει τις προσπαθίες του σε τέσσερα θέματα. Μεγαλύτερη ευαισθητοποίηση και ενημέρωση εντός της δίκησης, να βελτιωθεί η ανάλυση και παρακολούθηση και η διάδοση των πρόοδων στην πολιτική συνοχή, να βελτιωθεί η συνεργασία ε, μεταξύ των πρωταγωνιστών στο πλαίσιο των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, αυτή τη στιγμή η Ισπανία αναπτύσσει ένα σχέδιο εταιρική κοινωνικής ευθύνης, λαμβάνοντας υπόψη τις κύριες διεθνείς συμφωνίες. Αυτό προκύπτει από την ανακοίνωση της Κομισιόν για την εταιρική κοινωνική ευθύνη που εγκρίθηκε τον Οκτώβριο του 2011, που παροτρύνει τα κράτη-μέλη να στραφούν προς αυτή την κατεύθυνση. Επίσης, το Μάρτιο του 2011 είχαμε την πράξη της ε, αηφόρου οικονομία όπου εκεί διπρόθεταν η εταιρική κοινωνική ευθύνη. και συμπεριλαμβάνεται η εντολή τη κυβέρνηση να θεσπίσει δείκτε για την αξιολόγηση τη εταιρική κοινωνική ευθύνη και να ενημερώσει σχετικά σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα. Γι' αυτό δημιουργήθηκε μια ομάδα εργασίας που αποτελείται από κρατικούς συμβούλους. Η Ισπανία επίσης ε, σεβέστηκε τις ε, αρχές του ΩΣΑ ε, για τα πρότυπα που πρέπει να διέπουν την εταιρική κοινωνική ευθύνη και το Υπουργείο, το Υπουργείο Εξωτερικών προωθεί σήμερα το σεβασμό των δικαιωμάτων από την πλευρά των επιχειρήσεων για την ανάπτυξη εταιρική κοινωνική ευθύνη στην περίοδο 2011-2014. Είναι πάρα πολύ ενοχλητικό αυτό, λέει ο πρόεδρο. Ε, να πούμε στην τεχνική υπηρεσία που κάνει αυτές τις δοκιμές να σταματήσει αυτό το πείραμα γιατί μας παρακολουθεί στο έργο μα. Μιλάμε για συνοχή της, πολιτι... της πολιτικής. Ε, βλέπετε εδώ πως δεν υπάρχει συνοχή. Αν ήταν αδιαίθουσα δεν υπήρχε πρόβλημα, αλλά συνεχίστε, πρέπει και να ολοκληρώσετε. Έχω χάσει και χρόνο, το λαμβάνετε υπόψη. Λοιπόν, ε, θεωρούμε ότι είναι πολύ, πολύ σημαντική η συμμετοχή του ιδιωτικού σημαίου στη συνεργασία, όπως αντικατοπτρίζεται στο τέταρτο σχέδιο. να τονίσω τη σημασία του έργου που υλοποιείται στην επιστηστική ασφάλεια. Η Σχετική Επιτροπή των Ηνωμένων Εθνών, η πιο συμμετοχική πλατφόρμα των Ηνωμένων Εθνών για την επιστηστική ασφάλεια, ξεκίνησε μία διαβούλευση για δύο χρόνια για να αναπτύξει τις αρχές για υπεύθυνες αγροτικές επενδύσεις. Εκεί πρέπει να λαμβάνονται υπόψη όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη έτσι ώστε να έχουμε αηφόρες επενδύσεις που να συνεισφέρουν στην ανάπτυξη. Δημιουργήσαμε μια πυρική οπάδα για καλύτερη συνοχή μεταξύ ισπανικών και διεθνών πολιτικών. Αυτό το έργο θα συνεισφέρει επίσης στη θεματική διαβούλευση για το θέμα της πείνας και της διατροφής. Αυτή η διαβούλευση, μία από τις 11 που οργάνωσαν τα Ηνωμένα Έθνη στα πλαίσια της στρατηγικής για το 2015, είχε πολύ θετικά αποτελέσματα γιατί εστιάστηκε σε πολιτικές και τις παρουσίασε σε ένα έγγραφο που θα αποτελέσει τη βάση για τις εργασίες της Γενικής Συνέλευσης το Σεπτέμβριο του 2013. Για να ολοκληρώσω, η συνοχή είναι ένα στόχο ε, που σημαίνει ότι πρέπει να θέτουμε μακροπρόθεσμου στόχου και επομένω πρέπει να οικοδομηθεί μια πολιτική συνένεση για ε, να διατηρήσουμε τι υποσχέσει μα. Και πέρα από ότι προοδευτικά θέτουμε την συνοχή στη στρατηγική μα, είναι πάρα πολύ πιο δύσκολο να τεθεί σε εφαρμογή. Γι' αυτό ε, σύμφωνα με το όσο το Συμβούλιο στις 14 Μαρτίου, θα θέλαμε να έχουμε ένα μηχανισμό συνεργασίας και εφαρμογή ε, των αρχών αυτών μεταξύ κρατών μελών και Ευρωπαϊκής Ένωσης, κυρίως να ενισχύσουμε το διάλογο μεταξύ των Εθνικών Κοινοβουλίων και των κρατών μελών με τα Ηνωμένα Έθνη και τον ΟΗΕ, τον ΟΗΕ και τον ΟΣΑ και την ε, κοινωνία των πολιτών, έτσι ώστε να έχουμε καλύτερη αποτελεσματικότητα στις προσπαθίες μας. Σας ευχαριστώ Πρόεδρε. Και εγώ ευχαριστώ και στο συγγνώμη για όλες αυτές τις ε, ε, παρεμβάσεις οι οποίες, ε, όλες αυτές τις διακοπές που έγιναν. Προχωρώ τώρα στην Ουγγαρία και ζητώ να πάρει θέση ο εκπρόσωπος ή εκπρόσωπος της Ουγγρικής Βουλής για το θέμα της συνοχής. Ευχαριστώ Πρόεδρε και πριν ξαναρχίσει τώρα ο συναγερμός να πω πολύ γρήγορα ότι έχω και καλές ειδήσει και κακές ειδήσει. Αυτή τη στιγμή δεν ε, έχει η Ουγγρική κυβέρνηση αναπτυξιακή στρατηγική. Σήμερα το πρωί όμως ε, ε, το Υπουργείο Εξωτερικών στην Ουγγαρία φτιάχνει το πρώτο προσχέδιο μιας τέτοιας στρατηγικής. Από εκεί και πέρα όμως υπάρχουν πολλοί μη κυβερνητικοί οργανισμοί και γίνεται και η στρογγυλή τράπεζα η αυτών των μη κυβερνητικών οργανισμών η οποία κατέληξε συγκεκριμένες συστάσεις. Ήδη από το 2011 το κόμμα των Πρασίνων ε, που, το, που εκπροσωπώ κατάφερε να επιτύχει συνένεση μεταξύ πέντε κομμάτων και το Κοινοβούλιο ενέκρινε ψήφισμα το οποίο ζητεί από το Υπουργείο Εξωτερικών να φτιαχτεί μία ε, αναπτυξιακή στρατηγική για συνεργασία και σε περιφερειακό και σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Όταν έγινε η συζήτηση εκείνη στο Κοινοβούλιο, εγώ είπα ότι θα πρέπει να αναθεωρηθούν και να εξειδικευθούν λίγο παραπάνω οι τρέχουσες πολιτικές για να είμαστε σίγουροι για την αποτελεσματικότητα των προγραμμάτων αυτή τη στιγμή δεν δίνονται μεγάλα ποσά αλλά έχουμε διαπιστώσει ότι και αυτά τα μικρά ποσά ε, τα οποία διατίθενται ε, θα μπορούσαν να έχουν καλύτερα αποτελέσματα αν υπήρχε στενότερη συνεργασία καλύτερος συντονισμός και με γειτονικέ χώρες ε, εμείς μιλάμε τώρα για ποσά Φαίνω ύψους μισού εκατομμυρίου ε, ευρώ τα ποσά είναι πάρα πολύ μικρά όπως είπα και από εκεί και πέρα πρέπει να υπάρχει συντονισμός μεταξύ των διαφόρων υπουργείων Βεβαίω, υπάρχουν οι χώρες του Βίσεγκρατ που θα μπορούσαν να συνεργαστούν μεταξύ τους με, με κυβερνητικοί οργανισμοί αυτών των χωρών ενώ εν πάση περιπτώσει οι βουλευτέ των τεσσάρων χωρών ε, συναντήθηκαν και συζήτησαν θέματα αναπτυξιακή βοήθειας σε χώρες δεν είναι βέβαιος τυχαίο ότι οι περισσότεροι ο μεγαλύτερος και μη κυβερνητικό οργανισμός μεταξύ αυτών των χωρών είναι το People in Need που είναι τσέχικος οργανισμός θέλουμε ε, να, να ενισχυθούν και προσπάθειες άλλων οργανισμών σε αυτές τις τέσσερις χώρες ε, γίνονται προσπάθειες τις οποίες τις ε, μελετήσαμε γιατί υπήρχαν έργα στην Αιθιοπία και στην Κένια πριν από δύο χρόνια ε, από, βεβαίως οι Τσέχοι έχουν ε, μεγαλύτερη εμπειρία, ε, βοηθούν τις άλλες τρεις χώρες και εγώ προσωπικά επιμένω και προσπαθώ ότι ένα παράδειγμα βέλτιστης της πρακτικής είναι αυτό ακριβώ που κάνουν οι Τσέχοι. Το θέμα λοιπόν δεν είναι μοναχά να αυξήσουμε τα ποσά τα οποία διατίθεται για αναπτυξιακή βοήθεια, αλλά να προσπαθούμε προσπαθήσουμε να ε, ε, συνεργαστούμε, να συντονιστούμε για να έχουν καλύτερη απόδοση αυτά τα χρήματα. Θα πρέπει να οργανωθούν σωστά οι προσπάθειες και βεβαίως και εμείς σαν πρέπει να εξασφαλίσουμε ότι τη λογοδοσία για τα χρήματα αυτά και πρέπει να επιλέξουμε τις βέλτισες πρακτικές τις οποίες θα πρέπει να προσπαθήσουμε να επιβάλλουμε. Ε, χαίρομαι, είμαι αισιόδοξη, νομίζω ότι υπάρχει ένα μέλλον σε αυτές τις προσπάθειες. Ευχαριστώ Είναι εκπρόσωπο του Γκρικού Κοινοβουλίου. Θα δώσω τώρα το λόγο στον εκπρόσωπο του Κοινοβουλίου της Πορτογαλίας στην εκπρόσωπο. Ευχαριστώ, καλημέρα σας. Ε, θα έχει δύο μέρη η παρέμβασή μου θα σα αναφέρω και ποιε πολιτικέ. βρίσκουμε στην Πορτογαλία και τι ε, πρωτοβουλίε που έχει θετήσει το κοινοβουλίο μα. Μια πιο αξιοπρεπή ζωή για όλου είναι το τελικό σκοπό όλων των αναπτυξιακών πολιτικών να εγγυθούμε ότι όλοι οι άνθρωποι θα ζουν σε ελευθερές συνθήκε, χωρί φόβο και ε, χωρί ε, ανάγκε εδώ. Θέλουμε να εγγυηθούμε την αποτελεσματική των αναπτυξιακών πολιτικών. Ο αντίκτυπος των αποφασιών μας σημαίνει ότι θα έχουμε παγκόσμια δικαιοσύνη, σεβασμό ανθρώπινων δικαιωμάτων και περισσότερη ασφάλεια. Και εμεί σε αυτό το πλαίσιο κινούμαστε. Η συνοχή τη αναπτυξιακή πολιτική πρέπει να έχει συγκεκριμένο επιχειρησιακό περιεχόμενο. Η συνοχή σημαίνει διάρθρωση και σημαίνει ότι πρέπει να έχουμε συνέργειες, πρέπει να αποφύγουμε τις επικαλύψεις και ε, πρέπει να προωθούμε την αηφόρο ανάπτυξη. Δεν ε, πρέπει ε, βέβαια να ξεχνάμε το πλαίσιο στο οποίο βρισκόμαστε. Σημερινά μερινά σενάρια συρρήκνωση των προπολογισμών να αντιμετωπίσουμε όλοι πάρα πολλέ οικονομικέ δυσκολίε και ε, πρέπει οι εξωτερικέ πολιτικέ να είναι περισσότερο συνεκτικές. Η καλύτερη συνοχή των εθνικών πολιτικών προ την αναπτυξιακή πολιτική είναι κάτι θεμελιώδε για την αποτελεσματικότητα της ε, ε, πολιτικής της Πορτογαλίας. Η Πορτογαλία ε, προσυπογράφει τη συνοχή της αναπτυξιακής πολιτικής ε, σύμφωνα με τις ε, δεσμεύσεις που έχουμε αναλάβει είτε στην Ευρωπαϊκή Ένωση είτε στα Ηνωμένα Εθνή είτε στον ΕΣΑ. Τον Οκτώβριο του 2010 η Πορτογαλία ήταν σε ένα κατάλογο τεσσάρων μόλις χωρών που είχαν τέτοια νομοθεσία. Έτσι λοιπόν θεωρούμε ότι οι πολιτικές που έχουν υιοθετηθεί σε διάφορες τομές να συνάδουν με τους αναπτυξιακούς στόχους απόφαση του Συμβουλίου των Υπουργών να αναγνωρίζει το να έχουμε τους κατάλληλους μηχανισμούς συντονισμού προκειμένου να ενισχυθεί ο διυπουργικός διάλογος με συστηματικό και αποτελεσματικό τρόπο. Γι' αυτό συστήσαμε μια ομάδα εργασία για το θέμα αυτό κατόπιν ενός προγράμματος από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή 2010-2013 ενισχύουμε ε, τις πιο σχετικές πολιτικές για την επίτευξη των στόχων της ε, χιλιετίας όπως είναι αλλαγή, το εμπόριο, επιστημική ασφάλεια, μετανάστευση και ασφάλεια. Αυτό μα επιτρέπει επίση να αναγνωρίσουμε ότι από την εθνική σκοπιά έχουν αναπτυχθεί μηχανισμοί συντονισμού επικαιροποιημένοι, δημιουργήθηκαν συνέργειε προκειμένου να αυξηθεί η αποτελεσματικότητα των εθνικών πορτογαλικών πολιτικών. Και στο πλαίσιο αυτό εγκρίθηκαν στην Πορτογαλία διάφορα στρατηγικά έγγραφα που συνδέουν τι διάφορε τομεκέ πολιτικέ και θέλουν καλύτερη συνοχή μεταξύ στόχων και αποτελεσμάτων, όπω η Εθνική Στρατηγική για την ε, ε, ε, ασφαλή, για την ανάπτυξη στα πλαίσια ασφάλεια η Πορτογαλία υιοθέτησε και ένα ψήφισμα για την ασφάλεια της ανάπτυξης και εκεί όπως είπε η Χίλερη Μπάν, ε, η υπουργό αρμόδια για την εξωτερική ανάπτυξη, δεν είναι δυνατόν ε, να έχουμε ασφάλεια χωρίς ε, ανάπτυξη και η ασφάλεια χωρίς ανάπτυξη είναι μόνο εφήμερη. Επομένως, σε ό,τι αφορά τώρα τις πρωτοβουλίες των Ευρωπαϊκών του Πορτογαλικού Κοινοβουλίου έχει λάβει διάφορες ε, μορφές. Ε, καταρχήν έχουμε μια καθημερινή πρακτική στις ε, νομοθετικές μου πρωτοβουλίες. Ο κάθε βουλευτής ε, ξέρει ότι ε, η δουλειά του σε κάθε επιτροπή μπορεί να προωθήσει το έργο άλλων επιτροπών, αλλά μπορεί και να το υποσκάψει. Ε, όταν μιλάμε για τη συνεργασία στην υγεία, πρέπει να λάβουμε υπόψη την κοινωνική πρόνοια, τη γεωργία, την παιδεία. Τώρα προετοιμάζουμε μια βασική νομοθεσία προκειμένου να συνδέσουμε τομεακές πολιτικές ε, που είναι σημαντικές για το μέλλον της χώρας, όπως παραδείγματο χάρη οι πολιτικές για το είδωρ. Και πρέπει ε, να δούμε πώς διαρθρώνονται η δράση των πολιτικών ε, ομάδων, των κοινοβουλευτικών ομάδων σε όλο αυτό. Ε, μία απόφαση που εθετήθηκε από το Κοινοβούλιο προτρέπει την κυβέρνηση να σεβαστεί τον τέταρτο και πέμπτο στόχο της χιλιετίας, δηλαδή να βελτιωθεί η υγεία ε, των ε, γυναικών, μητέρων και να μειωθεί η παιδική θνησιμότητα. Μία άλλη μορφή άσκησης ε, των αρμοδιοτήτων μας είναι ε, το να παρεμβαίνουμε στην Ολομέλεια. Έχουμε τοποθετηθεί υπέρ της συνοχής και επίσης ε, έχουμε θέσει και ερωτήσεις στους αρμόδιους υπουργούς επίσης. Υπάρχει και ένα project για την συνοχή των αναπτυξιακών πολιτικών και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και εκεί δόθηκε ένα στέρι, δηλαδή αναγνωρίστηκε ότι αποτελεί μια ε, καλή πρακτική. Επίσης έγινε μια ακρόαση με τους αρμόδιους υπουργούς για αυτούς τους φακέλους και αναφέρθηκε ότι η συναχή της ανεπτυξικής πολιτικής επιφέρει πρόσθετη αξία και υπάρχει πολιτική συνένεση. Να σας ε, τονίσω ότι υπάρχουν πάρα πολλές πρωτοβουλίες και πάρα πολλά σεμινάρια και δημόσιες πρωτοβουλίες. Ολοκληρώνω, λέω μιλήτρια. Έλεγα ότι είχαμε πάρα πολλά σεμινάρια και δημόσιες δράσεις που υλοποιήθηκαν στο Κοινοβούλιο. Επίσης, να πούμε ότι στις 14 Μαΐου θα έχουμε μία συνεδρίαση για τα ανθρώπινα δικαιώματα, για την ε, στρατηγική μετά το 2015. Ελπίσουμε η δική μας πρακτική να μπορέσει να τροφοδοτήσει τη συζήτηση και σας ευχαριστώ για τη συζήτηση αυτή. Ελπίζω να είναι υποοικοδομητική και να σας πω ότι εδώ προσπαθούμε να οικοδομήσουμε μια μεγαλύτερη αξιοπρέπεια ε, και η συνοχή της αναπτυξιακής πολιτικής είναι ένα πολύ σημαντικό τμήμα όλου αυτού του καθημήματος που προσπαθούμε να οικοδομήσουμε. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ. Δίνω το λόγο στον πρόσωπο του Ηνωμένου Βασιλείου. Εστέ σύντομος παρακαλώ. Ευχαριστώ. Όπως γνωρίζετε από το 1997 το Ηνωμένο Βασίλειο έχει ένα ξεχωριστό Υπουργείο ανεξάρτητο από το Υπουργείο Εξωτερικών και έχει και μια κοινή κοινοβουλευτική επιτροπή για την ανάπτυξη. Δύο παράγοντες πρέπει να ληφθούν υπόψη στη, για το Ηνωμένο Βασίλειο. Πρώτα πρώτα να πούμε ότι υπάρχει ε, ε, διακομματική απόφαση για το 0,7% και υπάρχει και η απόφαση ε, πιο πρακτικά για 11 και κάτι εκατομμύρια στερλίνες που είναι το 0,7%. Βεβαίως επικρίθηκαν οι αποφάσεις αυτές από τα ΜΜΕ, από την δεξιά πτέρυγα του Συντηρητικού Κόμματος και από το UKIP που όπως φαντάζομαι θα ξέρετε ε, όχι απλώς είναι κατά της ανάπτυξης αναπτυσσόμενης χώρες αλλά και κατά της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Παρόλα αυτά είμαστε είμαστε αποφασισμένοι να υποστηρίξουμε την ε, αναπτυξιακή βοήθεια και να εξασφαλίσουμε ότι κάνουμε πράγματα τα οποία αποδίδουν καρπούς. Βεβαίως για το θέμα της συνοχής υπάρχουν πολλά πράγματα που θα μπορούσαμε να πούμε. Η τωρινή κυβέρνηση έκανε μια αναθεώρηση της διμερούς και ε, πολυμερούς βοήθειας, μείωσε τον αριθμό των διμερών εταίρων από 45 σε 28 και επέκρινε και πολλές από τις αναπτυξιακές από τους αναπτυξιακούς οργανισμούς μη κυβερνητικούς οργανισμούς και γιατί δεν κατάφεραν να μειώσουν ε, το επίπεδο της φτώχειας που συνδέεται με την μη συνδεδεμένη βοήθεια ε, αλλά μπαίνει στο ίδιο ο, ε, κεφάλαιο αν θέλετε με την αναπτυξιακή βοήθεια που η σχέση βεβαίως με την Ευρωπαϊκή Ένωση ε, σε αυτή την ανασκόπηση, την αναθεώρηση ε, αναλύθηκε θετικά εκείνο που επικρίθηκε ε, είναι το ποσό τα παγκόσμια ταμεία ε, θεωρήθηκε ότι δρούν πάρα πολύ καλά ε, και σε εκείνες τις χώρες όπου το Ηνωμένο Βασίλειο έχει διμερεί προγράμματα ο πρόσωπος του Ηνωμένου Βασιλείου ε, θαρρύνει το συντονισμό μεταξύ των χορηγών βοήθειας και όταν η Επιτροπή μας πάει σε κάποια χώρα με την οποία έχουμε διμερή συνεργασία πάντα γίνεται μια ε, στρογγυλή τράπεζα με άλλους χορηγούς βοήθειας και έχουμε έτσι τους χορηγούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης, την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, την USAID, το Καναδά, την Ιαπωνία κτλ. Ε, και την Κίνα και γιατί προσπαθούμε να κινητοποιήσουμε τους Κινέζους σε σχέση με την Αφρική. Όμως εκείνο που πρέπει τώρα να πούμε είναι το εξή ότι καταφέραμε να φτάσουμε στο 0,7% το διατηρούμε, το εφαρμόζουμε. Αυτό είναι καλό. Όμως πρέπει να δουλέψουμε περισσότερο για είναι το συντονισμό και τη συνοχή. Και το DFID που είναι αρμόδιο για την ε, αναπτυξιακή βοήθεια προσπαθεί να κάνει ακριβώς αυτό. Θέλουμε στο, σύνοδο κορυφής του G8 να συζητηθούν θέματα φορολογικά. Δεν θα μπορούσαμε να βάλουμε και εκεί ένα κομμάτι στην, ε, που σχετίζεται με τα φορολογικά ε, που έχουν σχέση με την αναπτυξιακή και της χώρας. Αποδέκτες ανέφερα τα βιοκαύσιμα προηγούμενα στην ερώτησή μου. Ε, και είναι μεγάλο το πρόβλημα των βιοκαυσίμων και σχετίζεται βεβαίως με το τι κάνουμε γενικότερα στη Γεωργία. Ε, συμπέρασμα. Υποστηρίζουμε αυτά που έλεγε ο Επίτροπος προηγούμενα καταρχήν Χρειάζεται κοινό προγραμματισμό. Υπό ένα όρο όμω, πρέπει να είμαστε ρεαλιστικοί. Οι εθνικέ κυβερνήσει θα πρέπει να αναλάβουν τη δεσμεύση για, να, για την χορήγηση αναπτυξιακή βοήθεια. Βεβαίω υπάρχουν ιδιαιτερότητε και ο καθένα καθορίζει τη δική του αναπτυξιακή βοήθεια, αλλά θα πρέπει να συνεργάζονται οι εθνικέ κυβερνήσει με του άλλου χορηγού, ούτω ώστε να εξασφαλιστεί ότι πραγματικά οι χώρες τις οποίες δίνουμε τη βοήθεια αυτή ενστερνίζονται τις, ε, τους στόχους μας και έτσι θα αποδώσει η βοήθεια την οποία χορηγούμε. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ, Σερ Μπρούς. Ευχαριστούμε και τους συναδέλφους που παρουσίασαν παραδείγματα ε, για τις βέλτιστες πρακτικές. Ε, θα ήθελα τώρα να γίνει μια συζήτηση μεταξύ των α, παρευρισκομένων. Θα ήθελα να πείτε ποιοι είστε και από πού προέρχεστε. Πρώτη πρώτη η κυρία Αρένα ζητεί το λόγο. Βέλγιο νομίζω. Euh, ναι, από τη Βουλή. Από τη Γερουσία με συγχωρείτε. Τη Γερουσία. Σύμφωνο για την ανάγκη συνοχής και επίτευξη του 0,7%. Σίγουρα δεν θα αλλάξουμε έτσι τον κόσμο. Γι' αυτό θα με ενδιαφέρει περισσότερο το 50% το οποίο, από το οποίο αποφελούνται τελικώς οι ευρωπαϊκές χώρες. Μιλάω για την επιστηστική βοήθεια, για τα θέματα τα εμπορικά, για τη βοήθεια για το περιβάλλον κλπ. Σημαντικά θέματα επί των οποίων πρέπει να συντονιστούμε. Έχουμε επίσης τις συμφωνίες ελευθέρων συναλλαγών, ε, θέματα προστασίας επενδύσεων. Εμείς στη Γερουσία του Βελγίου έγιναμε ψήφισμα το οποίο υπευθύνουμε και στην Ευρωπαϊκή Ένωση, όπου λέμε ότι πρέπει σε όλε τι συμφωνίε ελευθέρων συναλλαγών και για την προστασία των επενδύσεων πρέπει να υπάρχει μια ρήτρα κοινωνική και περιβάλλοντο, η οποία θα διατυπώνεται ρητό και η οποία θα προβλέπει και κυρώσει στην περίπτωση μη συμμόρφωση, ώστε να προφυλάσσεται η κυριαρχία των τρίτων χωρών. Θέλουμε λοιπόν σε κάθε περίπτωση να προστατεύσουμε την κυριαρχία των κρατών. Μετά, διαφάνεια για του προπολογισμού. Μιλήσαμε για διαφάνεια όσον αφορά του κρατικού προπολογισμού και εννοείται ότι είμαστε υπέρ προκειμένου, αλλά ζητούμε να υπάρχει διαφάνεια και όσον αφορά την εσωτερική λογιστική των πολυεθνικών. Υπάρχει μια ευρωπαϊκή πρωτοβουλία για το θέμα αυτό. Θέλουμε η οδηγία η σχετική να εφαρμοστεί και οι αρχέ του ΩΣΑ για την διαφάνεια να μην είναι αντικείμενο αλλά υποχρεωτικής συμμόρφωση όσον αφορά τις πολυεθνικές οι οποίες έχουν παρουσία στην επικράτεια της Ευρωπαϊκή Ένωση. Ευχαριστώ πολύ, ήσασταν και εξαιρετικά σύντομοι. Κύριος Άγγελ, Μαρκ Άγγελ Λουξεμβούργο. Πρόεδρε, αγαπητέ φίλε Σάγλ, μια λέξη για το τι κάνουμε για την συνοχή στο Λουξεμβούργο. Ξέρετε ότι εδώ και 10 χρόνια εμείς είμαστε πάνω από το 0,7%. Είμαστε ήδη στο 1% εδώ και δύο χρόνια του ΑΕΠ του Λουξεμβούργου και υπάρχει πολιτική συνένεση σε εθνικό επίπεδο μεταξύ κυβέρνηση και πολιτικών κομμάτων υπέρ αυτής της θέσης. Και αυτό παρά το γεγονός των δημοσιονομικών περιορισμών. Στο Λουξεμβούργο τροποποιήσαμε τον νόμο για την συνεργασία εγώ υπέβαλα πρόταση το 2009 ώστε η λέξη συνοχή να ενσωματωθεί στην νομοθεσία μας. Με την κυβέρνηση λοιπόν καταρτήσαμε και θεσπίσαμε νόμο στον οποίο δύο άρθρα αφορούν τη συνοχή των πολιτικών. Στο άρθρο 6 συγκεκριμένα λέμε ότι κάθε χρόνο ο Υπουργός υποβάλλει έκθεση για την πολιτική ανάπτυξη στη Βουλή προφορικός και γραπτός και ένα κεφάλαιο αφορά συγκεκριμένα τη συνοχή των πολιτικών. Επίσης, δημιουργήσαμε Διπουργική Επιτροπή για την συνεργασία με σκοπό την ανάπτυξη, γιατί εκπροσωπούνται όλα τα Υπουργεία και συσκέπτονται τακτικώς για να συζητήσουμε θέματα ανάπτυξης. Η συνοχή λοιπόν είναι κατοχυρωμένη δια νόμου, αν και δεν έχει υλοποιηθεί πλήρως, γι' αυτό και οι προσπάθειες συνεχίζονται. Τρίτον, σε εργασία μεταξύ Βουλής του Λουξεμβούρου και ΜΚΟ οι οποίες συναντώνται μάλιστα και με την Υπουργική Επιτροπή, πρέπει να πω. Μία φορά το χρόνο λοιπόν, στο πλαίσιο της σύσκεψης της ε, Επιτροπής Εξωτερικών ε, Σχέσεων, αποτυπώνουν την υλοποίηση των πολιτικών, με γνώμονα όλα αυτά για την καλύτερη εφαρμογή των πολιτικών, αλλά και η ενημέρωση της κοινή γνώμη, όχι μόνο μεταξύ κυβέρνηση φυσικά, ΜΚΟ και βουλευτών. Θέλουμε να δώσουμε αυτό το παράδειγμα λοιπόν Συνοχή στον τομέα των βιοκαυσίμων σχετικά με την αλλαγή του κλίματος κλπ. Έχουμε καταρτήσει επίσης ένα χρονοδιάγραμμα το οποίο προσπαθούμε να καταστήσουμε όσο και πιο συνακτικό γίνεται στη Βουλή, όσον αφορά τι συζητήσει δηλαδή με γνωμόνα με θέμα την ανάπτυξη. Κάθε χρόνο λοιπόν, κάθε Ιούλιο, ο Υπουργό, όπω είπα, υποβάλλει έκθεση στην Σχετική Επιτροπή. Τον Σεπτέμβριο μετά το Υπουργείο, μαζί με τη ΣΜΚΙΟ και τη Βουλή, επί τρίμερο, συνεδριάζουν για να συζητήσουν θέματα ανάπτυξη. Καλούμε πρέσβει, ε, ΜΚΙΟ, από τι χώρε αποδέκτε τη βοήθεια κλπ. Και, και τον Οκτώβριο, εν συνεχεία, έχουμε και την ετήσια συζήτηση για τα μετά συνεργασία με σκοπό την ανάπτυξη. Υπάρχει ένα ταμείο αποζημίωση το οποίο διαχειρίζεται χρήματα συνταξιδοτικών ταμείων. Ω τώρα τα ταμεία αυτά επενέβαιναν σε βιομηχανίε όπλων. Τώρα το ταμείο αυτό, το νέο αυτό ταμείο, επενδύει μόνο σε επιχειρήσεις οι οποίοι συμπεριφέρονται με τρόπο υπεύθυνο όσον αφορά το περιβάλλον και την κοινωνία. Προσπαθούμε επίση στον με των κρατικών προμηθειών, των δημοσίων συμβάσεων, να κάνουμε τα αντίστοιχα. Αυτά με δύο λόγια. Αν έχετε ερωτήσει, παρακαλώ στη διάθεσή σα. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ, Μάρκ Άγγελ. Θα έλεγα ότι δίνετε μακράν το καλό παράδειγμα ως χώρα. Και τώρα, κύριε Λίλη Τεσουές, ελπίζω να μην ε, προφέρω λάθος το όνομά σας. Καλημέρα. Λέγομαι Λίλι Βαλόντος. Εκ μέρους της Επιτροπής που εκπροσωπώ, την Επιτροπή Εξωτερικών Σχέσεων του Σουηδικού Κοινοβουλίου, ήταν από το εξή. Τα ερωτήματα αυτά είναι εξαιρετικά επίκαιρα και θέλω να Πω δύο λόγια σχετικά. Τρεις παρατηρήσεις θα ήθελα να καταθέσω συγκεκριμένα. Πρώτον, η Επιτροπή των Εξωτερικών Σχέσεων έλαβε πρωτοβουλία να συντάξει έκθεση σαν απόκριση της θέσης της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε διεθνείς διαπραγματεύσεις για το πλαίσιο μετά το 2015. Η θέση μας είναι ότι η εξάλληψη της φτώχειας και η φορεία συνδέουν μεταξύ τους. Συνεπώς, η δράση μας από εδώ και πέρα για τους στόχους της χιλιετίας και η ατζέντα για το 2020 πρέπει να συγκεραστούν. Δεύτερον, στον τομέα της αλληλείας, της γεωργίας, του περιβάλλοντος και του εμπορίου, μεταξύ άλλων βεβαίως, είναι φανερό ότι οι αποφάσει τη Ευρωπαϊκή Ένωση ε, επηρεάζουν τα μάλλα τη αναπτυσσόμενες χώρες. Και τέλο, λαμβάνουμε υπόψη μα τον ρόλο τη Ευρωπαϊκή Ένωση ω το μεγαλύτερο δωρητή στον κόσμο και τις δεσμεύσει φυσικά που έχουμε αναλάβει. Εν αυτών, η Επιτροπή θεωρεί ότι η αναπτυξιακή συνεργασία πρέπει να διδαματίσει κυρίαρχο ρόλο στο πλαίσιο μετά το 2015. Και αναμένω σχετικό στα σχολεία σας. Ευχαριστώ πολύ. Euh, σας ευχαριστώ. Και τώρα να δώσω το λόγο στον κύριο Πολσίνοβιτς από την Κροτία. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Είναι μεγάλη τιμή για μένα να εκπροσωπώ τη χώρα μου στη συζήτηση αυτή καθώς εμείς ε, πρόκειται να μπούμε στην Ευρωπαϊκή Ένωση σε δύο μήνες και σας ευχαριστώ για την ε, ευκαιρία που μας ε, δώσατε και εδώ αλλά και σε άλλους δεσμούς να αρχίσουμε να συνεισφέρουμε και εμείς στη χάραξη των σημαντικών πολιτικών. Θα ήθελα να δράξω την ευκαιρία για να σας πω ότι η Κροατία λόγω του μεγέθους της, είναι μια μικρή χώρα και έχοντας τους δικούς της στόχους ε, προσπαθεί να ακολουθήσει τις ε, κύριες αυτές που διέπουν την περιφερειακή ανάπτυξη. Έχουμε επικεντρωθεί σε δύο κυρίους τομείς. Καταρχήν θέλουμε να βοηθήσουμε τη δική μας περιφέρεια και ξέρετε αυτές τις μέρες έρχονται θετικά νέα από την περιοχή αναφέρομαι στη Συμφωνία Σερβίας Σερβίας-Κοσικοπεδίου και ε, Επίσης, ε, να συνεισφέρουμε με τη δική μας μοναδική εμπειρία στις διαπραγματεύσεις. Ξέρετε, διαπραγματευτήκαμε με ένα πολύ μοναδικό τρόπο και προσπαθούμε να διαβιβάσουμε τη γνώση που έχουμε αποκτήσει από αυτή τη διαδικασία σε άλλους εταίρους ε, της ε, ευρύτερης περιοχής στην Ανατολική Ευρώπη. Και έτσι έχουμε συστήσει ανακεντρωριστίες για τη διαβίβαση αυτής της γνώσης που είναι πολύ σημαντική για την ανάπτυξη της ε, περιοχής μας. Επίσης, συμμετέχουμε πάρα πολύ ενεργά στις διεθνείς αποστολές και επιχειρήσεις. Προσπαθούμε να συνδέσουμε αυτά τα δύο. Έχουμε παρουσία στο Αφγανιστάν από το 2003, το χάρη, και μέχρι τώρα έχουμε επενδύσει σε πάνω από 40 διαφορετικά προγράμματα, ακολουθώντας ε, τις κυρίες αρχές ε, της κοινή πολιτικής μας, ε, δηλαδή επενδύσεις στην υγεία, στην παιδεία, στην οικοδόμηση κτηρίων, κρατικών και την ανάπτυξη μικρών επιχειρήσεων. Πριν δύο ημέρες ανοίξαμε ένα νέο σχολείο στη τη Σαρίφ και ξεκινήσαμε μια μικρή επιχείρηση με γυναίκες που λέγεται Χαλιά από το Αφγανιστάν. Σας ευχαριστώ λοιπόν για την ευκαιρία αυτή και ανυπομονώ να είμαι και πλήρες μέλος, τακτικό μέλος ε, στις συνεδριάσεις ε, και στην συμμετοχή πολιτικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Πρόεδρος, ε, επειδή δεν έχουμε πολύ χρόνο, θα ολοκληρώσω τον κατάλογο, θα κλείσω τον κατάλογο των ομιλητών, θα δώσω το λόγο σε όσους μου τον έχουν ζητήσει μέχρι τώρα, αλλά δεν θα δεχτώ αιτήματα. Η κυρία Ρούτσιν από την Πούντερστακ, από την Κατούβουλη. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Πρώτα πρώτα θα ήθελα να ευχαριστήσω για την όλη συζήτηση. Είναι πρώτη φορά που κάνουμε μια τέτοια άτυπη συζήτηση. Ε, δείχνει ότι κερδίζει έδαφος όλο και, όλο και περισσότερο έδαφος η συνεργασία μεταξύ των Εθνικών Κοινοβουλίων. Αυτό είναι πάρα πολύ καλό γιατί μας βοηθάει να προσεγγίσουμε και τις, τρε, απόψεις μας για τη στρατηγική μας. Ε, θα ήθελα να συγχαρώ το Ηνωμένο Βασίλειο που έφτασε στο 0,7 του ΑΕΠ για την αναπτυξιακή βοήθεια. Εμείς δεν τα έχουμε καταφέρει, είμαστε στο 0,39 ακόμη βεβαίως πρόσφατα ε, και εμείς έχουμε ένα Υπουργείο Αρμόδιο για την Ανάπτυξη που ε, έχει αποκοπεί, είναι αυτόνομο σε σχέση με το Υπουργείο Εξωτερικών και ελπίζουμε ότι θα τα πάμε καλύτερα στο μέλλον. Γι' αυτό ακριβώς το λόγο. Από εκεί και πέρα όλες οι ευρωπαϊκές πρωτοβουλίες που σχετίζονται με την αναπτυξιακή όλες τις ευρωπαϊκές πρωτοβουλίες που σχετίζονται με την αναπτυξιακή πολιτική προσπαθούμε να τις ομαδοποιήσουμε και να τις συζητήσουμε ε, στην δική μας επιτροπή. Συζητήσαμε δηλαδή θέματα ας πούμε των ε, εμπορικών ε, συν συμφωνιών Κολούμπια Περού παραδείγματος χάρη δεν είχαμε όλοι τις ίδιες απόψεις είχαμε διαφορετικές απόψεις άρα τι θέλω να πω θέλω να πω ότι δεν προσπαθούμε να έχουμε συνοχή μόνο σε αυτά που κάνει η χώρα μας σε σχέση με την αναπτυξιακή βοήθεια αλλά προσπαθούμε να υπάρχει συνοχή και σε αυτά που γίνονται σε ευρωπαϊκό επίπεδο ε, προσπαθούμε να έχουμε μια κοινή θέση και αυτό προσπαθούμε να το μεταφέρουμε στις Βρυξέλλες. Αυτό θα πρέπει να διευρυνθεί περαιτέρω. Θα πρέπει να υπάρχει συνοχή και μεταξύ των Εθνικών Κοινοβουλίων και από εκεί και πέρα. Δεν λέω ότι θα πρέπει να κοροϊδευόμαστε και να αγνοούμε το γεγονός ότι υπάρχει πρόβλημα στα όσον αφορά τη συνοχή και το συντονισμό. Υπάρχουν προβλήματα, αλλά σαν βουλευτές θα πρέπει να φροντίσουμε τα θέματα τα οποία τίθεται σε ευρωπαϊκό επίπεδο ή σε άλλες χώρες να τα συζητούμε και να προσπαθούμε να τα συντονίσουμε γιατί αυτό δεν είναι καθόλου αυτονόητο αυτή τη στιγμή. Ευχαριστώ πολύ λέει ο πρόεδρος η κυρία Μπάγερ από την Αυστρία είναι η τελευταία ομιλήτρια. Ευχαριστώ πολύ. Να πω πρώτα πρώτα ότι εμείς στην Αυστρία ε, επιβάλλεται δια νόμου η αναπτυξιακή συνοχή η συνοχή στην αναπτυξιακή πολιτική. Βεβαίω, μην με ρωτήσετε πώς εφαρμόζεται, διότι δεν είμαστε και πολύ καλοί, δεν έχουμε καταφέρει να βρούμε εκείνα τα εργαλεία τα οποία μας ε, ε, βοηθούν να έχουμε με μεγάλο βαθμό συνοχής. Βεβαίως έχουν γίνει πρόοδοι στο κοινοβούλιο και πραγματικά εκείνο που βλέπουμε είναι να συναντιούνται οι βουλευτές μας που ασχολούνται με τα θέματα αυτά συχνά και να έχουν και πολύ συχνές επαφές με τους μη κυβερνητικού οργανισμούς. Αυτό είναι θετικό. Υπάρχει μια έκθεση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ε, του 2011 για την ε, συνοχή ευρωπαϊκής ε, αναπτυξιακής πολιτικής. Αυτό είναι αυτό που μας κάνει να οργανώνουμε αυτές τις αιτήσει συναντήσεις και αυτό είναι πολύ καλό και σε αυτή την έκθεση περιγράφονται πολύ καλά συγκεκριμένα μέτρα στην παράγραφο 21 συγκεκριμένα λέγεται ότι αυτή η δομημένη ε, συνάντηση θα πρέπει να ορίζει και στόχους οι οποίοι να είναι ελέγξιμοι. Αυτό το χαιρετίζω, αυτό είναι πάρα πολύ καλό, είναι πάρα πολύ συγκεκριμένο. Σας ρωτώ λοιπόν, υπάρχουν τέτοια μέτρα. Υπάρχουν μέτρα, υπάρχει ένα κατάλογο κριτηρίων που είχε λεχθεί ότι θα φτιαχτεί για να τα ελέγξουμε και για να μπορέσουμε να ξεκινήσουμε με βάση κάτι το πολύ συγκεκριμένο να δουλεύουμε. Ε, σαν βουλευτές νομίζω ότι μπορούμε να βοηθήσουμε σε αυτή την συνοχή των κοινωνικών πολιτών αναπτυξιακών πολιτικών και στο δικό μας στο καθένα στο δικό του κοινοβούλιο αλλά και στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και αν δεν υπάρχουν ακόμη τέτοια μέτρα ε, θα πρέπει να σκεφτούμε πολύ σοβαρά να τα αποφασίσουμε Σας ευχαριστώ. Φτάνουμε στο τέλος μιας πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση. Ε, ήταν πολύ ενδιαφέρουσα χάρη στι ε, διάφορες παρεμβάσει Σε αυτό το τμήμα τη συζήτηση. πήραν το λόγο μόνο μέλη των Εθνικών Κοινοβουλίων ε, οι Ευρωβουλευτέ, Σας άκουσαν πάρα πολύ προσεκτικά και μπορώ να σας εγγυηθώ ως μόνιμος εισηγητής για τη συνοχή της αναπτυξιακής πολιτικής. Σημείωσα τις προτάσεις σας και κυρίως ε, της τελευταίας πρότασης της κ. Μπάιερ. Το χρονοδιάγραμμα προβλέπει να παρουσιαστεί η έκθεση της Επιτροπής ε, του κ. Βίμπαλξ ε, μέχρι το Σεπτέμβριο. Κατόπιν το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα συνεχίσει τις εργασίες που έχουν ήδη ξεκινήσει ε, η Επιτροπή Ανάπτυξης μου έχει, θέσει μία, μου έχει αναθέσει μία εντολή με κάποια σημεία και θα πρέπει εγώ να δω πώς μπορούμε να βελτιώσουμε τις ε, πολιτικές συνοχής και φυσικά ε, με την ε, συμφωνία και με ε, τις ε, μη κυβερνητικέ οργανώσεις που δραστηριοποιούνται εδώ στις Βρυξέλλες και κάνουν πάρα πολύ σημαντική δουλειά. Θα ήθελα να σας δώσω λίγο χρόνο, αλλά δυστυχώς δεν μας περισσεύει και θα ήθελα να πω κάποια λόγια συμπερασματικά. Φυσικά θα πρέπει να καταρτήσουμε μία σειρά κριτηρίων έτσι ώστε να έχουμε μία κοινή εκτίμηση της κατάστασης σε σχέση με τη συνοχή των πολιτικών. Στον ΟΣΑ συνεχίζονται οι εργασίες, οι σχετικές, συμμετέχουμε και εμείς ως άτομα ή εκπροσωπώντας την Επιτροπή μας στις εργασίες αυτές. Θα πρέπει να έχουμε μια κοινή ανάγνωση, γιατί ο στόχος της συνοχής ε, των πολιτικών εγγράφεται στη συνθήκη της Λισαβόνας και θα πρέπει να αποκτήσουμε τα μέσα για να υλοποιήσουμε τα όσα λέγονται στη συνθήκη, τη διάταξη της συνθήκης. Ε, δεύτερον, αυτή η συνεδρίαση αποτελεί σε μια πολύ καλή ευκαιρία για να ανταλλάξουμε απόψεις σε θεμελιώδη ζητήματα. Στα εισαγωγικά μου σχόλια υπενθύμησα ότι η συνοχή των πολιτικών σημαίνει να σεβαστούμε όλα όσα έχουν οικοδομηθεί στους άλλους ε, τομείς. τομέα ε, της αναπτυξιακής συνεργασίας. Ε, ένας, ε, οι τομείς που ανταγωνίζονται το τομέα είναι τα βιοκαύσιμα, η κοινή αγροτική πολιτική δεν είναι ουδέτερη για το θέμα ε, του επισητισμού και των τροφίμων. Παγκοσμίως, επίσης θα πρέπει να δούμε και το θέμα της μεθόδου. Και θα ήθελα να κάνω κάποια σχόλια από αυτού εδώ, στο ιστορικό του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Είδατε ότι υπήρξαν κάποιες δυσκολίες για να ξεκινήσει η διαδικασία εποπτείας ε, της συνοχής των πολιτικών στις χώρες σας και το ίδιο συνέβη και στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Δεν ε, νομίζω ότι σα αποκαλύπτω κανένα κρατικό μυστικό, λέγοντας ότι εδώ στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο πολλές φορές έχουμε δυσκολίες ε, να συζητήσουμε με τις υπόλοιπε επιτροπές. Ε, θα πρέπει να γίνει κάτι τέτοιο, χρειάζεται μια παιδαγωγική προσέγγιση και φυσικά θα πρέπει να λάβουμε και κάποια μέτρα για να καταλήξουμε εκεί. Η κατάσταση τώρα δεν είναι ικανοποιητική κατά την άποψή μου. Και Φυσικά πρέπει να σεβαστούμε το καθεστώς των επιτροπών στο ιστορικό αυτό του Κοινοβουλίου που αποτελεί και μια διεπαφή ανταλλαγή απόψεων με τους άλλους εταίρους και είναι σημαντικό αυτό να ανταλλάσσουμε απόψη με τους υπόλοιπους ε, κοινοβουλευτικούς εταίρους. Είμαστε 28 πρωταγωνιστές που πρέπει να συνηθούν για τον έλεγχο αυτής της αναπτυξιακής πολιτικής και δεν είναι εύκολο να αναλάβουμε τον έλεγχο αυτό. Γιατί δεν ε, εντάσσονται τα αποτελέσματα στον προϋπολογισμό ε, και ε, ξέρετε ότι τα κράτη-μέλη αποφασίζουν το μέγεθος του προϋπολογισμού και ο ρόλος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου είναι πολύ περιορισμένος γιατί δεν συμπεριλαμβάνεται στη συνθήκη. Έτσι λοιπόν πώς θα πράξουμε έτσι ώστε όλοι να έχουν μία κοινή εκτίμηση έτσι ώστε και οι 28 ε, να συγκλίνουν προς ε, τις ε, απαιτούμενες κοινέ δράσεις στα πλαίσια της αναπτυξιακής συνεργασίας. Τι θα μπορούσαμε να κάνουμε για να βελτιώσουμε την κατάσταση. Θα σας κάνω μια πολύ απλή πρόταση. Εγώ είμαι υπεύθυνο για τη σύνταξη αυτή τη έκθεση. Εκπροσωπείτε τα Εθνικά Κοινοβούλια. Μην διστάσετε να απευθυνθείτε στη γραμματεία μα με τι δικέ σα προτάσει, τι προσδοκίε σα και σας προτείνω ότι από τη στιγμή που ε, θα υπάρχει η πρώτη εκδοχή της ε, Έκθεση αυτή σας προτείνω να σας τη στείλω. Μην διστάσετε λοιπόν να χρησιμοποιήσετε αυτή τη δυνατότητα και εγώ θα σας ευχαριστούσα για κάτι τέτοιο, θα σας ήμουν ευγνώμων. Και κατόπιν ε, και ο κ. Μισελ, ο οποίος είναι συντονιστή ε, του ΕΛΚΟΔΑ στην Επιτροπή Ανάπτυξης, ε, σίγουρα θα συμφωνεί μαζί μου ότι πρέπει να επαναλάβουμε αυτή την εμπειρία. Και εγώ, αν χρειαστεί, μπορώ να έρθω να σας επισκεφτώ στα εθνικά σας κοινοβούλια για να συζητήσουμε τα θέματα αυτά της συνοχής της αναπτυξιακής πολιτικής. Μέσα από την ποικιλομορφία ε, των ε, απόψεων σας είδαμε ότι έχουμε ένα μακρύ δρόμο να διανύσουμε για να συγκλίνουν οι μέθοδοι εργασίας μας και οι απόψεις μας. Για να αναφέρω ένα παράδειγμα, έχουμε δύο προσεγγίσεις που μου φαίνονται παραδειγματικές. Αν θυμάμαι καλά, η πρώτη αφορά μια συνήθεια που δημιουργήθηκε στο Συμβουλίο των Υπουργών ε, στις κάτω χώρες. Ε, σε κάθε συνεδρίαση του Υπουργικού Συμβουλίου υπήρχε από το υπεύθυνο της αναπτυξιακής συνεργασίας μία ενημέρωση. Και να, αυτό είναι συνοχή των πολιτικών. Και ένα δεύτερο παράδειγμα που θα μπορούσα, από το οποίο θα μπορούσα να μα εμπνεύσει είναι κάτι που ανέφερε η κυρία Ρότ από την Bundestag. Αναφερθήκατε στη δική σα επιτροπή που επίση γνωμοδοτεί για το τι κάνουν οι στο τομείς που αφορούν την αναπτυξή συνεργασία περισσότερο ή λιγότερο. Αυτό είναι ένα παράδειγμα σε ό,τι αφορά τώρα το στόχο του, το στόχο του 0,7% είμαι σίγουρος ότι είστε κινητηρίως δύναμη, ότι δίνετε πολιτική όφηση σε αυτό το ζήτημα τα αποτελέσματα είναι πάνω κάτω μη ικανοποιητικά. Υπάρχουν α, κάποιες χώρες και χάρηκα πολύ άκουσα τον πρόσωπο του που μας είπε ότι ό,τι και να γίνει Εμεί θα φτάσουμε στο 0,7%. Και αυτό είναι πολύ σημαντική πολιτική επιλογή. Δεν μπορούμε να σα υποστηρίξουμε σε αυτό το θέμα. Και κάτι που μου φαίνεται πολύ σημαντικό είναι ότι κατορθώσατε αυτό να ε, το πετύχετε ε, παρά ε, τις πολιτικές διαφωνίες. Σας ευχαριστώ λοιπόν πάρα πολύ. Ξέρω και τι λένε διαφορετική σε σχέση με το 0,7%. Λοιπόν, ε, υπήρχε και αυτή μικρή δυσκολία, οι τεχνικές υπηρεσίες δυσκόλεψαν τις εργασίες μας. Όμως παρόλα αυτά η ποιότητα των παρεμβάσεων σας ε, ήταν πολύ ικανοποιητική και ευχαριστώ και τον συνάδελφο ε, Μίτσελ, Μίτσελ. Θα του δώσω το λόγο. Δεν ξέρω τι πρόκειται να σας πει, αυτό θα σας τα παρουσιάσει. Σας δίνω το λόγο. Ευχαριστώ. Thank you. Um, First, let me thank you for your presence at this interparliamentary meeting. Να σας ευχαριστήσω. Και η Μίτσελ είναι το όνομά μου, μέλος και συντονιστής της Επιτροπής Ανάπτυξης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και εισηγητής της νομοθετικής πρωτοβουλίας για τον συντονισμό των δωρητών στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Χαίρομαι που μαζευτήκαμε εδώ σήμερα, χάρη στην Προεδρία η οποία έστειλε τον Πατ Μπριν εδώ πρόεδρο της αντίστοιχης επιτροπής ε, της ε, Ελληνικής Βουλής. Μιλούμε λοιπόν για τον συντονισμό των ε, αναπτυξιακών πολιτικών. Θα μιλήσουμε για συνοχή μεταξύ ευρωπαϊκών πολιτικών. Μιλήσαμε μάλλον γι' αυτό. Τώρα θα μιλήσουμε για τον συντονισμό των αναπτυξιακών πολιτικών. Μιλήσαμε για τη βοήθεια λοιπόν. Τώρα θα μιλήσουμε για την ανάπτυξη. Ο συντονισμό των δωρητών πρέπει να αποτελέσει ένα συνεκτικό πλαίσιο την επιτεύξη των στόχων της ανάπτυξης. Η συνοχή εν προκειμένου αφορά πολιτικές σε διάφορους τομείς εκτός από την ανάπτυξη αυτή καθ' Πρέπει καταρχήν να φροντίσουμε ότι η μία πρωτοβουλία δεν υποσκάπτει την άλλη. Το ζήτημα της καλύτερης του καλύτερου μάλλον συντονισμού προϋποθέτει συγκεκριμένου χειρισμού και απάντηση στο ρώτημα πώς πρέπει να χορηγείται η βοήθεια. Πώς θα αντιμετωπίσουμε το θέμα του κατακαιρματισμού ή του κατατομέα κατακαιρματισμού της βοήθειας. Πώς θα πετύχουμε λοιπόν με αυτά που έχουμε τα καλύτερα αποτελέσματα. Για κάθε δηλαδή ευρώ που πληρώνει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Ο συντονισμό των δωρητών είναι ουσιαστικά η διαδικασία στο πλαίσιο τη οποία οι χώρε συνεργάζονται για την βελτιστοποίηση τη απόδοση. Παρ' όλα αυτά, ο συντονισμό δεν είναι αυτό σκοπό. Αυτό που μα ενδιαφέρει είναι το τελικό αποτέλεσμα. Το θέμα είναι να περιορίσουμε μεταξύ άλλων τις, ε, τα χρηματοπιστωτικά έξοδα για να κάνουμε περισσότερα με τη συγκεκριμένη επένδυση. Αυτό απαιτείται πολύ περισσότερο σήμερα εν ώψη της ε, ακραίας λιτότητας σε πολλές ευρωπαϊκές χώρες, κατά το οποίο απομειώνει την παρέμβαση, τη σημασία της παρέμβασης της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Είμαστε ο μεγαλύτερος δωρητής. Πρέπει ως μεγαλύτερος δωρητή, η Ευρωπαϊκή Ένωση και τα κρατημέλη να φροντίσουν η βοήθεια αυτή να χορηγείται αποτελεσματικά. Οι δομέ που έχουμε στη διάθεσή μα, μα επιτρέπει να συγκρίνουμε, να μαθαίνουμε, να καταγράφουμε τι καλύτερε πρακτικέ και να τι εφαρμόζουμε. Αν ρίξουμε μια ματιά γύρω μας όμως, θα δούμε ότι αυτό δεν συμβαίνει πάντα. Ο αντίκτυπος της ε, βοήθειας που χορηγούμε είναι μικρότερο από αυτόν που θα έπρεπε. Διότι σπαταλούμε πόρους, πολλοί το ονομάζουν αυτό το κόστος της Ευρώπης. Με άλλα λόγια, εμείς που ζούμε εδώ στην Ευρώπη, Πρέπει να ξέρετε ότι δίνουμε περισσότερη από τη μισή βοήθεια που δίνεται ανά τον πλανήτη και όμως αυτή δεν αποδίδει πάντα. Το αμήλικτο γεγονός είναι ότι κάθε μέρα πεθαίνουν 23.000 παιδιά σε όλο τον κόσμο. 23.000 παιδιά σήμερα, αύριο και μεθαύριο. Θα πρέπει να τα μειώσουμε στο μισό. Επίσης, στον αναπτυσμένο κόσμο η παιδική θνησιμότητα είναι 68 της χιλής. 68 της χιλής. Μην ξεχνάτε ότι στην Ελλανδία και σε άλλες χώρες μετά τον, στο τέλος του Δεύτερου Παγκοσμίου Πολέμου ήταν 48. Εκεί φτάσαμε. Στον αναπτυσμένο κόσμο είμαστε στο 63 σήμερα έναντι 2013. Δεν είναι μόνο θέμα ανθρωπιστικό. Επίσης μην ξεχνάτε ότι το 2050 θα έχουμε 2 δισεκατομμύρια πλέον πληθυσμό στον ε, πλανήτη. Γι' αυτό τα παιδιά πρέπει να κάνουμε κάτι. Χρειάζεται λοιπόν καλύτερη εξελόγηση των πολιτικών, Χρειάζεται καλύτερο συντονισμό. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο αυτή τη στιγμή διερευνά αυτό το κόστο. Το κόστο τη μη Ευρώπη, όπω το ονομάζουμε, και τη έλλειψη συντονισμού. Η Επιτροπή Ανάπτυξη παρήγγειλε αυτή τη μελέτη, η οποία οριστικοποιήθηκε και δημοσιεύθηκε τον Ιούνιο του 2012. Εκεί επιβεβαιώνεται ότι ο συντονισμό θα αποφέρει μόνο φελήματα. 800 εκατομμύρια ευρώ θα μπορούσαμε να περισσώσουμε κάθε χρόνο ως Ευρωπαϊκή Ένωση μόνο και μόνο από την απομείωση την, τον, τον περιορισμό του χρηματοοικονομικού κόστους και του κόστους των συναλλαγών, του κόστος της διαδικασίας. Αυτή η εξοικονόμηση θα μπορούσε να απελευθερώσει περισσότερα κονδύλια ακριβώς υπέρ των αναπτυσσομένων χωρών. Ο καλύτερος συντονισμός θα σημάνει επίση υψηλότερη αποτελεσματικότητα, καλύτερη παρακολούθηση, περισσότερη διαφάνεια. Άρα και καλύτερα αποτελέσματα. Η εναρμόνιση επίση έχει ωφελήματα και για τις ε, χώρε αποδέκτες. Λιγότερα διαδικαστικά κόστη, υψηλότερη απορρόφηση και καλύτερη διακυβέρνηση. Από πολιτικής απόψεως, ο συντονισμό και η εναρμόνιση θα συμβάλλουν στην επίτευξη των στόχο μας και θα επιτρέψουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση να ελοπίσει την φιλοδοξία της να παραμείνει ένας πρωταγωνιστής στο διεθνέ προσκήνιο. Ο στόχο του 0,7% για το 2015 παραμένει ένα μακρινό στόχο για τι περισσότερε χώρε. Παρά τι αξιόπαινε πρωτοβουλίε του Ηνωμένου Βασιλείου. Αν και κάποιοι κατηγορούν το Ηνωμένο Βασιλείου την έλλειψη υποστήριξη. Και όμω υπάρχουν ευρετανικέ προσπάθειε που αποτελούν πολύ καλό παράδειγμα. Για άλλη μια φορά, απαιτείται καλύτερο συντονισμό. Όπω ε, έδειξε η έρευνα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, η επικέντρωση λιγότερε χώρε και σε πιο συγκεκριμένε δραστηριότητε είναι εκ των νουκάνευ. Αυτό θα διευκολύνει την προσπάθεια καλύτερου συντονισμού στο πλαίσιο και της ε, Εκρήξης άκρα των Μπουσάν και των Παρισιών. Θα συνεχίσουμε λοιπόν να συνεργαζόμαστε στενότερα σε ευρωπαϊκό επίπεδο για καλύτερη κατανομή εργασιών στο πλαίσιο ενός κοινού προγράμματος. Στην πράξη έχουμε δει σε πολλές περιπτώσεις ότι αυτές οι βασικές αρχές όμως εναπόκεινται, επαφίενται στον πατριωτισμό, όπως λέμε, των των μελών και σε διμερή συντονισμό. Εν γέννη, Όλοι οι φορεί που παρέχουν βοήθεια συμφωνούν ότι απαιτείται καλύτερο συνερισμό. Στην πράξη όμω τα πράγματα δεν είναι τόσο απλά. Τα κράτη-μέλη έχουν το καθένα την άποψή του για το τι πρέπει να γίνει. Αλλά δεν δείχνουν και τόσο έτοιμα να κάνουν συμβασμού. Επίση, η προσπάθεια καλύτερου συνερισμού συνεπάγεται και πολιτικό κόστο για κάποιε χώρε που θα φαίνονται λιγότερο, αν θέλετε, ω δωρητές. Αλλά και αυτό θα μπορούσαμε να το λύσουμε. Ίσως μια χώρα δωρητής να είναι επικεφαλής μιας ευρωπαϊκής προσπάθειας και εκεί να φαίνονται όλοι. Από το 2010 εμείς το Συμβούλιο και στην είπατε εκπρόσωπο και τις υπηρεσίες της δημιουργήσαμε νέες θέσεις για την ανάπτυξη και τη βοήθεια. Αυτό όμω έχει και κινδύνους. Χρειάζεται λοιπόν περαιτέρω συζήτηση και προσοχή. Καλό είναι να τονίζουμε τα κέρδη από τον καλύτερο συντονισμό στο μέλλον, αλλά το θέμα είναι να βρούμε και τα συγκεκριμένα εργαλεία για το πώς θα το κάνουμε αυτό, πώς θα αναπτύξουμε δηλαδή τον συγκεκριμένο συντονισμό και όλα αυτά να πάρουν τη μορφή μια νομοθετική πρωτοβουλία του Κοινοβουλίου. Ω συζητητή τη συγκεκριμένη πρωτοβουλία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, σκοπεύω να προτείνω και περαιτέρω νομοθετήματα τα οποία θα κάνουν πιο απτά τα ωφελήματα από τον καλύτερο συντονισμό. τη συνάδελφη αναγνωρίζω, αντιλαμβάνομαι τον κρίσιμο ρόλο των εθνικών κοινοβουλίων. 26 χρόνια ήμουν μέλο ενό εθνικού κοινοβουλίου και γνωρίζω πολύ καλά πόσο κρίσιμη σημασία είναι η συμβολή των Εθνικών Κοινοβουλίων. Γι' αυτό άλλωστε βρισκόμαστε και εδώ σήμερα. Εκφράζω λοιπόν την ικανοποίησή μου και τον ενθουσιασμό μου για τη σημερινή συζήτηση και προσβλέπω στις ε, απόψει. Απαντήσει στα ερωτήματα Πώ θα πετύχουμε καλύτερο συντονισμό των αναπτυξιακών πολιτικών τη Ένωση και των κρατών μελών. Ποιο είναι ο ρόλο των Εθνικών Κοινοβουλίων, του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Πώ θα πείσουμε τι κυβερνήσει να συμφωνήσουν και να γίνουν υπόλογε στα Εθνικά Κοινοβούλια και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Εμεί ω Εθνικά Κοινοβούλια δεν θέλουμε να υποκαταστήσουμε φυσικά το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στον ρόλο του. Το θέμα είναι τι θα κάνουμε μαζί. Πόσο σημαντική μετά είναι η μείωση του μη παραγωγικού κόστου χάρη στο συντονισμό. Τέλο, ε, πώ θα επικεντρώσουμε του δωρητέ στα βραχυπρόθεσμα αποτελέσματα. Πώ θα σταματήσουμε να σπαταλούμε τη βοήθεια. Και πώς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και τα Εθνικά Κοινοβούλια θα διασφαλίσουν ότι η εξοικονόμηση πόρων θα πάει τελικώς στις αναπτυγμένες χώρες με καλύτερη απόδοση. Επιτρέψτε μου να δώσω τον λόγο στον κύριο Κρυμό, ο οποίος είναι επικεφαλής ε, της ε, μονάδας μας στη Γενική Διεύθυνση ΔΕΦΚΟ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Ε, Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Κυρίες και κύριοι βουλευτές, θα ήθελα να παρουσιάσω πολύ σύντομα ορισμένα πράγματα σχετικά με το συντονισμό των χορηγών βοήθειας. Αυτό είναι κλασικό θέμα με το οποίο ασχολούμεθα και νομίζω ότι σήμερα είναι πολύ σημαντικό, ακόμη πιο σημαντικό σήμερα, γιατί έχουμε δύο προκλήσεις να αντιμετωπίσουμε. Από τη μια έχουμε τη διεύρυνση και από την άλλη έχουμε την εμβάθυνση. Ε, διεύρυνση. Εδώ και δεκαετίες ε, συντονίζονται οι χορηγοί βοήθειας μέσω διαφόρων μηχανισμών. Από την άλλη μεριά όλο και καινούργιοι παίκτες μπαίνουν στην αγορά των δωρητών. Η Κίνα παραδείγματος χάρη, οι αραβικές χώρες ε, και άρα η πρόκληση είναι αυτή η πρόκληση της διεύρυνσης του αριθμού αν θέλετε των περισσότερων χορηγών και το πώς αυτοί θα ενταχθούν σε ένα σύστημα συντονισμένο. Όταν ε, το 2011 έγινε το φόρουμ για την αποδοτικότητα και την αποτελεσματικότητα της βοήθειας. Αυτό ακριβώς ήταν ένα θέμα που συζητήθηκε για τις αναδυόμενες χώρες, τους καινούριους δωρητές κτλ. Από Πρέπει λοιπόν να εμπλακούν και οι νέες αυτές χώρες με, τις, με τους εταίρους μας. Είναι σημαντικό το πρόβλημα, ε, δεν λέω ότι είναι αδύνατο να γίνει, αλλά πρέπει να φροντίσουμε γιατί όσο περισσότερο εντάσσονται και οι νέες αυτές χώρες τόσο μεγιστοποιείται ή το αποτέλεσμα της βοήθειας. Δεύτερη πρόκληση που ανέφερε ήταν η ευάθυνση. Τι θα πει αυτό. Ο συντονισμός σε ευρωπαϊκό επίπεδο, Ευρωπαϊκή Ένωση, κράτη-μέλη ας πούμε. Αυτός υπάρχει εδώ και κάμποσα χρόνια. Όμως, άμα δούμε την πραγματικότητα τι γίνεται με τη βοήθεια βλέπουμε έναν κατακαιρματισμό όπως είπε ο κύριος Μίτσελ της βοήθειας αυτής οι Ευρωπαίοι χορηγοί λοιπόν ε, είναι ε, κάνουν πράγματα είναι μέρος του προβλήματος. Υπάρχουν πολλοί χορηγοί Ευρωπαίοι που παρεμβαίνουν σε πολλούς και διαφορετικούς τομείς κατακαιρματίζεται λοιπόν η βοήθεια τα χρήματα του Ευρωπαίου φορολογουμένου τα οποία δεν αποδίδουν τους καρπούς που έπρεπε να αποδώσουν εδώ και αρκετά χρόνια βεβαίως έχουν παρθεί πρωτοβουλίες για να ενισχυθεί περισσότερο ο συντονισμός μεταξύ των Ευρωπαίων χορηγών. Μπορώ να σας δώσω πάρα πολλά παραδείγματα για αυτά που γίνανε από το 2010 και δόθε. Ε, θα αναφέρω δύο. Το 2004 ε, ο κώδικας δεοντολογίας για την ε, ε, κατανομή εργα... καθηκόντων εργασίας μεταξύ των διαφόρων χορηγών και διαφόρων τομέων. Αυτή τώρα όμως η πρωτοβουλία του 2007 τώρα αντιμετωπίζει δυσκολίες γιατί θα πρέπει να παρέμει κανείς αυτό σε ένα συγκεκριμένο στάδιο όπου παίρνονται οι αποφάσεις και γι' αυτό καταλήξαμε τώρα στον κοινό προγραμματισμό συζητήθηκαν τα θέματα αυτά σας λέω στο φόρουμ του Μπουσάν ε, και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή επιμένει ακριβώς όπως μας είπε και ο Επίτροπος προηγούμενα στο κοινό προγραμματισμό και σε κάτι τι άλλο θέλουμε σε κάποιες χώρες να γίνονται κοινέ αναλύσεις κοινέ αναλύσεις μεταξύ Ευρωπαϊκών Ευρωπαίων χορηγών για να γίνεται και κατανομή α, αρμοδιοτήτων για να μην υπάρχουν επικαλύψεις για να υπάρχουν τα μέγιστα πιθανά αποτελέσματα. Είναι δύσκολα τα πράγματα αλλά αν καταφέρουμε να υπάρχει συντονισμός και κατανομή σωστή των διαφόρων ε, στους διάφορους χορηγών για τους διάφορους τομείς τότε το κέρδος θα είναι τεράστιο Επίσης θα είναι πολύ καλό αυτό και για την παρουσία των Ευρωπαίων χορηγών, την ορατότητά τους αν θέλετε και για τη δυνατότητα προ, ε, πρόβλεψης ορισμένων αναγκών για το μέλλον. Βεβαίω, τα διάφορα κράτη-μέλη, τα διά, διάφοροι εθνικοί οργανισμοί, τα εθνικά κοινοβούλια έχουν τι δικές τους προτεραιότητε. Θα πρέπει όμω να προσπαθήσουμε να τα συντονίσουμε όλα αυτά. Το άλλο το οποίο είναι πολύ σημαντικό είναι η αποκέντρωση. Ε, γιατί αποσυγκέντρωση αν μπορώ να το πω έτσι γιατί ορισμένα πράγματα αποφασίζονται σε διάφορες χώρες θα μπορούσαν να αποφασίζονται σε διάφορες πρεσβείες που έρχονται σε επαφή μεταξύ τους από εκεί και πέρα υπάρχει και ένα άλλο θέμα εφόσον θα είναι ο συντονισμό όσον αφορά το χρονοδιάγραμμα. Γιατί εφόσον υπάρχουν εθνικά σχέδια και εθνικά χρονοδιαγράμματα, εκεί θα μπορούσαμε να πέμβουμε Άλλο θέμα. Η Ευρωπαϊκή Ένωση και τα κράτη-μέλη είναι οι κύριοι ε, ε, ήδη έχουν ξεκινήσει την ιδέα αυτή του κοινού προγραμματισμού αλλά εκείνο που είναι σημαντικό είναι να πείσουμε και άλλους χορηγούς να ε, συνεργαστούν μεταξύ μαζί μας για να υπάρχει κοινό προγραμματισμός και με αυτούς. Να πω επίσης ότι όλες αυτές οι πρωτοβουλίες είναι και προαιρετικές και βαθμιές ε, ξεκινήσαμε με 7 χώρες και τώρα ε, έχουν προσθεθεί γύρω στις 30 ακόμη χώρες που λαμβάνουν μέρος αυτόν τον κοινό προγραμματισμό με τους οποίους προσπαθούμε να συγχρονιστούμε και περιμένουμε και άλλους όπως είπα. Αυτή τη στιγμή λοιπόν κυρίες και κύριοι έχουν γίνει ορισμένα πράγματα προσπαθούμε να προωθήσουμε όλες αυτές τις πρωτοβουλίες ε, είναι πολύ νωρίς για να δούμε κατά πόσον υπάρχει ικανή ε, πολιτική βούληση πίσω από όλα αυτά αλλά είναι πολύ σημαντικό όλοι να προχωρήσουμε και όπως είπε και ο κύριος Μισελ πρόσφατα η μεταξύ μας είμαστε όλοι ίσοι σε ευρωπαϊκό επίπεδο ως χορηγοί εκείνο που είναι σημαντικό είναι να συνειδητοποιήσουμε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι ο πρώτος και μεγαλύτερος χορηγός στον κόσμο και να δουλέψουμε όλοι μαζί για να αποδώσει καρπούς αυτή η δουλειά Σας ευχαριστώ τώρα μπορούν να συνεισφέρουν ε, και τα μέλη των κοινοβουλίων ε, ο κύριος Κάσπαρ καταρχήν. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ και Τσάρλς ε, για την ε, προηγούμενη παρουσίαση. Σήμερα είναι τα γενέθλια του Σέξπιρ. Αλλά θα πω κάτι από τον Όσκαρ Βάιλτ, ότι η αδερφότητα είναι ε, πολύ σημαντική δική του Άρους και ελπίζω να μπορέσω να το αποδείξω στη λογοδοσία. Λοιπόν, μάλλον, αν δούμε πώς ε, θα υπάρχει λογοδοσία σε εθνικά κοινοβούλια πρέπει όλες αυτές οι διαδικασίες να γίνονται δημόσια και κατόπιν οι βουλευτές ε, στις συνεδριάσεις των Εθνικών Κοινοβουλίων ε, να κάνουν τους υπουργού να λογοδοτήσουν ε, για το τι γίνεται. Επίσης πρέπει και οι χορηγοί της βοήθειας αλλά και οι δικαιούχοι να είναι κύριοι των project. Επίσης πρέπει να μειώσουμε το κόστος γιατί ο κίνδυνος είναι ότι αν δεν μειώσουμε το κόστος θα χάσουμε την αποτελεσματικότητα ποιότητα της βοήθειας και τέλος, και αυτό είναι μία έκκληση για τους συναδέλφους από τα Εθνικά Κοινοβούλια. Μπορείτε παραδείγματο χάρη να επιμείνετε στην αρχή ότι τα ανθρώπινα δικαιώματα είναι στο κέντρο των πολιτικών μας και δεν υπάρχει αποδυνάμωση αυτής της αρχής όταν προβαίνουμε σε μεγαλύτερο συντονισμό γιατί πολύ συχνά έχουμε σύγκρουση των πολιτικών όταν ε, το εμπόριο ουσιαστικά υπερισχύει τη αρχής του σεβασμού των ανθρώπων δικαιωμάτων. Αρικά πολύ που αναφερθήκατε στον συμπατριώτη μου Δουβλινέζο συγγραφέα. Στο... Στο έγγραφο του Ρίου Συνήκωση αναφέρονται ε, αρκετοί ότι στην ε, βιώσιμη ανάπτυξη και ότι ορισμένα πράγματα δεν έγιναν αλλά έκτοτε είδαμε ότι ότι ε, έχουν γίνει έκτοτε πολλά και έχουν συν, και συνεργάζονται κοινοβούλια, εθνικά κοινοβούλια μεταξύ τους. Πολλές χώρες και όπως και η δική μου μπο, ε, προσπαθούν να, τονί, να, να, προχωρήσουν όλα αυτά τα οποία αναφερθήκατε μεταξύ Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και Εθνικών Κοινοβουλίων είναι απαραίτητο να υπάρχει έντονη συνεργασία. Αυτή τη στιγμή ακόμη βέβαια δεν έχουμε κάποια θεσμική δομές που να ενισχύουν τη συνεργασία αυτή αλλά δεν σημαίνει ε, τίποτε ε, νομίζω ότι μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε άτυπες διαδικασίες έχουμε τηλεπικοινωνίες έχουμε τηλεδιασκέψεις έχουμε τέτοιου είδους μέσα που μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε για να συνεργαστούμε μεταξύ μας αυτό πρέπει να το τονίσουμε τα κοινοβούλια τα οποία είναι πολύ σημαντικά για την εφαρμογή ορισμένων πραγμάτων παραδείγματο χάρη στο Νότο ε, και που έπρεπε να έρθουν σε επαφή είτε με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο είτε με τα Κοινοβούλια του Βορρά χρησιμοποίησαν ορισμένα τέτοια μέσα. Δεν λέω ότι είναι πλήρης ότι υπάρχουν πολλά τέτοιου είδου μέσα αλλά θα πρέπει να τα ενισχύσουμε θα πρέπει να προσπαθήσουμε άτυπ, αυτές τις άτυπες μορφές επικοινωνίας να τις χρησιμοποιήσουμε για να μπορέσουμε να εστιάσουμε τη δουλειά μας και αργότερα φαντάζομαι ότι θα μπορούμε να προχωρήσουμε σε πιο επίσημες διαδικασίες, πιο θεσμικές δομές. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ, ο κύριος Λουμισελ. Ναι, καταρχήν συγχαρητήρια για την παρέμβασή σας, φυσικά την προσυπογράφουμε θα κάνω κάποιες συγκεκριμένες παρατηρήσεις. Καταρχήν, ε, συμφωνώ απόλυτα με την πρόταση του Μάικλ Κάσμαν να ανοίξουμε τις πόρτες μας στους εκπροσώπους ε, ε, των Εθνικών Κοινοβουλίων Ενωμένων Ομιλητής για τις, του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για τις τακτικές μας συνεργασίες. Δεύτερον, ίσως ε, θα ήταν ενδιαφέρον σε κάθε χώρα να υπάρχει ένας Ευρωπαίος συντονιστής που θα μπορούσε είτε να είναι κάποιο εκπρόσωπο τη Ευρωπαϊκή Ένωση είτε κάποιο ε, πρεσβευτής κράτους μέλου. Γιατί φυσικά θα μπορούσαμε να κατανείμουμε έτσι την εργασία για να υπάρχει πραγματικός συντονισμός σε κάθε χώρα Τώρα, το κόστος ε, της μη Ευρώπης. Κύριε Μίτσελ, εγώ πιστεύω ότι τα αριθμητικά στοιχεία που αναφέρετε δεν ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα, γιατί ε, τελευταία είδαμε ότι υπάρχει κατασπατάληση μέσων ε, για τα 49 το ευρώ που ε, εκταμιεύτηκαν από την Ευρωπαϊκή Ένωση, αυτό αποτελούσε ε, τελικά ένα ποσό που αντιστοιχούσε στα 6 έως 8 εκατομμύρια ετησίω. γιατί εκατομμύρια ετησίως, γιατί υπήρχαν ε, επικαλύψεις και υπήρχαν τεράστιες απώλειες. Έτσι λοιπόν χαίρομαι να έχω το αποτελέσμα αυτή της νέας μελέτης. Επίσης, Είμαι πεπισμένος ότι για να έχουμε ένα καλύτερο συντονισμό θα έπρεπε να στηριχθούμε περισσότερο στην εξειδίκευση των διάφορων χορηγών βοήθειας. Δηλαδή, πολλοί χορηγοί σήμερα κάνουν ε, το ίδιο πράγμα και όλα. Έτσι λοιπόν, παραδείγματο χάρη, ίσω θα έπρεπε να υπάρχει κάποιο κράτο μέλο, η Βρετανία, η Σουηδία ή το Λουξεμβούργιο. Αυτέ οι χώρε έχουν πραγματικά εμπειρία στι βελτιστέ πρακτικέ σε συγκεκριμένου τομεί. Μήπω θα έπρεπε λοιπόν να δούμε λίγο περισσότερο αυτό το θέμα τη εξειδίκευση. Επίση θα ήθελα να προσεγγίσουμε όχι σε επίπεδο συντονισμού, αλλά σε επίπεδο αποτελεσματικότητας της βοήθειας ε, να προσεγγίσουμε τα θέματα αυτά και να δούμε ποια είναι τα πλεονεκτήματα της ε, γενικής ε, δημοσιονομικής βοήθειας και της τομεακής γιατί υπάρχει το θέμα της ε, ευάλωτης κατάστασης ε, των κρατών και δεν μπορούμε να ενισχύσουμε τα κράτη παρά αν μέσα ε, αν διαθέσουμε μέσα στα κράτη αυτά για να πληρώσουν τους εκπαιδευτικούς, τους αστυνομικούς και γιατί αναφέρομαι σε αυτό, γιατί στα εθνικά μας κοινοβούλια συχνά υπάρχει μία ε, ε, εντύπωση κάπως αρνητική για την ε, δημοσιονομική βοήθεια και την τομεακή δημοσιονομική βοήθεια ότι δηλαδή δεν μπορούμε να ελέγξουμε τη χρήση της. Αυτό δεν ισχύει. Συστηματικά ελέγχεται η δημοσιονομική βοήθεια και μπορούμε να το κάνουμε και με τη βοήθεια του ελεγκτικού συνεδρίου. Ναι. Αυτό το θέμα για τα 800 εκατομμυρία ήταν ε, κόστος συναλλαγής. Εσύ αναφέρθηκες σε 6 δισεκατομμύρια, αλλά αυτό καλύπτει το σύνολο, ενώ εγώ αναφέρθηκα στο κόστος των συναλλαγών. Κύριε Χούμπνερ. Ευχαριστώ πολύ για τις παρεμβάσεις σας που ήταν πολύ ενδιαφέρουσες το Γερμανικό Κοινοβούλιο, η Γερμανική Κάτω Βουλή έχει ε, επανειλημμένα έρθει σε επαφή και με την Κομισιόν και έχει συζητήσει συναφή θέματα. Ε, γενικώ συμφωνούμε, αλλά πιστεύουμε ότι υπάρχουν συγκεκριμένα άλλα θέματα, όπως παραδείγματος χάνει εξειδίκευση που θα μπορούσαμε να συζητήσουμε. Είναι αυτό που είπε ο κύριο Μισελ. όταν έχουμε μία συνεργασία και όταν θέλουμε να καταλήμουμε καθήκοντα θα πρέπει να λάβουμε υπόψη την πείρα του άλλου γιατί ορισμένα κράτη-μέλη έχουν ειδικά εξειδικευθεί σε ορισμένα πράγματα και έχουν πολύ μεγάλη πείρα για σε ορισμένους τομείς. Ωστόσο υπάρχει κι άλλο ένα πρόβλημα και το είπαμε και στους υπουργούς μας και στο Υπουργικό Συμβούλιο ότι θα μια καλύτερη κατανομή καθηκόντων θα πρέπει να γίνει μεταξύ Ευρώπης γενικά Ευρωπαϊκής Ένωσης αφενός και κρατών μελών αφετέρου εδώ δεν υπήρχαν σαφή όρια στο παρελθόν και αυτό ήταν κακό για όλους όλοι αισθανόμαστε υπεύθυνοι για όλα αυτό δεν μπορεί να συνεχιστεί στο μέλλον θέλαμε λοιπόν να τονίσουμε ότι ειδικά η Ευρωπαϊκή Ένωση με τις ε, με τα, τι, τις δυνάμεις που έχει και τις γνώσεις που έχει για την αναπτυξιακή βοήθεια μπορεί να κάνει ορισμένα πράγματα και από εκεί και πέρα τα επιμέρους κράτη-μέλη θα μπορούσαν να δράσουν συμπληρωματικά ανάλογα με την πείρα του το καθένα. Σας ευχαριστώ, δεν βλέπω να ζητά άλλο το λόγο. Τότε να δώσουμε το λόγο στον εκπρόσωπο, το Φίλιξ Φερνάντες, ο προέρχεται από την ε, Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης. Πρόεδρε, ευχαριστώ που μας καλέσατε. Ό,τι είπε ο κ. Ε, Κρυμός, από την Κομισιόν, βεβαίως ε, ισχύει, συμφωνούμε. Συνεργαζόμαστε άλλωστε για τους σκοπούς του συντονισμού και του κοινού προγραμματισμού. Εν συντομία, δύο πράγματα που πρέπει επίσης να λάβουμε υπόψη μας ως προς τον συντονισμό. Εν γέννη συμφωνούμε σχετικά με τα περί αποτελεσματικότητας, ε, αντικτύπου, θέσπισης προτεραιοτήτων στις αναπτυσσόμενες χώρες κλπ. Και ότι όλα αυτά πρέπει να τα κάνουμε μαζί. Παρ' όλα αυτά, είμαστε ένας μεγάλος οργανισμός, εμείς εδώ στην Κομισιόν, στην υπηρεσία μας, τα 27 κρατημέλη, 28 κρατημέλη. Όλα αυτά λοιπόν πρέπει να μεταφραστούν σε συγκεκριμένες ε, δράσεις, σε συνεργασία με ΜΚΟ, με πρεσβείες και ούτω καθεξής. Εννοείται λοιπόν ότι εν γέννη απαιτείται καλύτερος συντονισμός στα πήκη κομισιόν. Πώς όλοι αυτοί οι φορείς σε επίπεδο χώρα, πρεσβείας, υπηρεσίες κλπ. Πώς θα εμπλακούν ταυτόχρονα στον ίδιο χώρο με το καλύτερο αποτέλεσμα όπως είπε και ο συνάδελφος, έχει σημασία πρώτον να συγχρονιστούμε. Δηλαδή να δουλεύουμε για τα ίδια θέματα ταυτόχρονα στον ίδιο χώρο. Αλλιώς, ο καθένας θα παίρνει τις αποφάσεις του σε διαφορετικά σημεία με αντικείμενο την ίδια χώρα. Και αυτό είναι πρόβλημα για τον προγραμματισμό και τον συντονισμό. Δεύτερον, να τονίσω ότι, όπως είπατε και εσείς κύριε Πρόεδρε, Υπάρχει μια θεσμική αλλαγή μετά τη Λισαβόνα. Το οποίο σημαίνει ότι οι αντιπροσωπείε τη Ευρωπαϊκή Ένωση έχουν διαφορετικό ρόλο πλέον. Έχουν αυτό που έκαναν παλιά, αλλά έχουν και έναν ρόλο συντονισμού των κρατών μελών όταν δρούν εκτό Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτό είναι σημαντικό βήμα, σημαντική πρόοδο για όλου μα, διότι υπάρχει εν τέλει συντονιστή επιτόπου, ο οποίο θα βάλει μια τάξη σε κράτη-μέλη και σε άλλους φορείς ή και σε μη Ευρωπαίους δωρητές. Γι' αυτό και ο Επιτροπός και ο κύριος Γκριμό είπαν ακριβώς αυτό, ότι μπορούμε να προγραμματίσουμε από κοινού σε επίπεδο χώρας λήπτη. Γι' αυτό εμείς, η Κομισιόν, ο Ευρωπαίος Φορολογούμενος, πληρώνουν διπλωμάτες και ειδικού επί θεμάτων ανάπτυξης για να δουλεύουν εκεί, στην περιοχή, στην Μπουρκίνα Φάσο, στην Βολιβία, στη Βολιβία ή αλλού, για να είναι εκεί, να γνωρίζουν τη χώρα και να ξέρουν τι πρέπει να γίνει. Αυτοί είναι σε θέση να πάρουν τις καλύτερες αποφάσεις, υποστηρίζοντας την Ευρωπαϊκή Ένωση όταν υλοποιεί αναπτυξιακή βοήθεια. Ας βασιστούμε λοιπόν στις αντιπροσωπείες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στην πρεσβεία μας, που θα συνεργαστούν φυσικά με τις πρεσβείες και άλλους φορείς αναπτυξιακής βοήθειας. Αυτό είναι μια καινούργια ιστορία, είναι μια καινούργια διαδικασία, ομολογώ, αλλά ήδη έχουμε τα πρώτα σημάδια επιτυχία. Ας ε, στηρίξουν τα κρατημέλη αυτήν την ε, διαδικασία που όπως είπα θα πρέπει να καταλήξει ένα κοινό προγραμματισμό. Μάλιστα από κοινού και με μη κοινωτικού δωρητέ, όπως είπε και ο Επίτροπο σήμερα το πρωί. Υπάρχει μια κοινή στρατηγική για την Αιθιοπία. Έχουν συνυπογράψει όλε οι χώρε, οι πρέσβεί και η κυβέρνηση τη Αιθιοπία. Υπάρχει συνεργασία. Να λοιπόν ένα καλό παράδειγμα που πρέπει να μιμηθούμε στο μέλλον. Όλα αυτά θα απαιτήσουν φυσικά χρόνο, διότι τα κράτη-μέλη και η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι μεγάλοι ογκώδεις ε, μηχανισμοί, υπάρχει μια κατανομή εργασία, υπάρχουν ένα σωρό πράγματα που πρέπει να ρυθμίσουμε θα γίνουν, αλλά πρέπει να γίνουν στο επίπεδο της χώρας λήπτη, ώστε η βοήθεια να είναι στοχευμένη. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ κύριε Φεράντες. Κότσε, παρακαλώ, κυρία. Ευχαριστώ πολύ. Η συνοχή είναι ένα θέμα για το οποίο χρειάζεται κυρίως ένα πράγμα, η πολιτική βούληση. Ρωτώ λοιπόν, διαπιστώνετε ότι υπάρχει πολιτική βούληση συνεργασίας, διότι αν δεν υπάρχει οι προσπάθειες που καταβάλουμε όλοι μας ή που συζητούμε ότι πρέπει να καταβάλουμε ε, είναι καταδικασμένες να αποτύχουν. Ρωτώ λοιπόν, Πού ανακαλύπτεται την πολιτική βούληση στις εθνικές κυβερνήσεις. Υπάρχει προθυμία. Αυτή η νοοτροπία σιλό και στεγανών που, ανα, που, ανα, που διαπιστώνεται στις διάφορες χώρες να αλλάξει. Και πιστεύετε ο, και ποια πιστεύετε ότι είναι η βούληση να προωθηθεί η αναπτυξιακή πολιτική σε σχέση με τις άλλες πολιτικές της διάφορες κυβερνήσεις. Εγώ πιστεύω ότι θα πρέπει από τη βάση, από κάτω να προκύψουν ορισμένα πράγματα στο εσωτερικό των κυβερνήσεων, στο εσωτερικό των κοινοβουλίων. Θα πρέπει να γίνει δουλειά ούτω ώστε από τη βάση να ξεκινήσουν κάποιες πρωτοβουλίες οι οποίες να προχωρήσουν μετά ομαδικά. Επανέργομαι στο βασικό ερώτημα. Υπάρχει πολιτική βούληση. Πού βρίσκεται αυτή η πολιτική βούληση ή μήπως η τάση είναι προς την αντίθετη κατεύθυνση. Μίτσελ, ευχαριστώ πολύ για την πολύ ενδιαφέρουσα ερώτηση. Εδώ είναι ακριβώς το κλειδί της υπόθεσης. Πώς θα διαλύσουμε αυτά τα στεγανά, αυτά τα σιλό που αναφέρατε. Εδώ πρόκειται για δημόσιο χρήμα, για το χρήμα των φορολογουμένων που πρέπει να διαπανάτε ε, με σοφρόνησίνη αλλά αποτελεσματικά. Ή, ήμουνα εισηγητής για την τον κανονισμό για επίγουσα βοήθεια ε, στις αρχές του καλοκαιριού φεύγαμε για διακοπές και το Σεπτέμβρη πήγα στη Γαλλία για να κάνουμε τη σχετική συζήτηση και γύρω στους 20-25 υπουργού μου είπαν ότι δεν θα μπορούσε να γίνει κάτι τέτοιο. Τελικά έγινε όμως εντός 100 ημερών. βρήκαμε τα χρήματα ε, και πέρασε η νομοθετική πράξη. Αυτό το λέω σαν παράδειγμα για το ότι ενώ δεν πιστεύουμε ότι ορισμένα πράγματα μπορούν να γίνουν, τελικά μπορούν να γίνουν. Ή μάλλον το πω αλλιώ. Στην Ιρλανδία το Ντόλ και η Γερουσία ε, μπορούν να περάσουν οποιαδήποτε νομοθετική πράξη θέλουν εφόσον δεν είναι αντίθετη προς το Σύνταγμα. Στο, στην Ευρώπη οι Ευρωβουλευτές δρούν διαφορετικά. Η ευρωβουλευτής λοιπόν δεν μπορεί να κάνει τη δουλειά του εθνικού βουλευτή ούτε το αντίθετο. Ε, πρέπει εμείς εδώ να σεβόμαστε το ρόλο του ημέν τον δε και να δούμε πώς μπορούμε να συνεργαστούμε. Είναι πολύ σημαντικός ο ρόλος των εθνικών κοινοβουλίων. Γι' αυτό έχουμε και αυτή, κάνουμε αυτή τη συνάντηση σήμερα ε, πρέπει να σεβόμαστε τα εθνικά κοινοβούλια αλλά και τα εθνικά κοινοβούλια πρέπει να σέβονται το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και να μπορούμε να συνεργαστούμε. Θεωρώ ότι είναι πραγματικά αξιοθαύμαστο ότι παρά τα προβλήματα που υπάρχουν στο Ηνωμένο Βασίλειο και λόγω και παρά όλη την κρίση που υπάρχει στην Ευρώπη το, το... το Ηνωμένο Βασίλειο πήρε διακομματικά την απόφαση για το 0,7%. Να λοιπόν ένα παράδειγμα για το ότι γίνονται ορισμένα πράγματα που δεν περιμέναμε να γίνουν. Βρισκόμαστε στην αρχή μιας διαδικασίας. Η έκθεση είναι ένα ρευστό έγγραφο. Θα συμπληρωθεί αργότερα το, το καλοκαίρι, το Σεπτέμβρη και ελπίζουμε και τα μέχρι τότε και τα, ευρωπαϊκά, τα εθνικά με συγχωρείτε κοινοβούλια να έχουν αποκρισταλώσει άποψη, να έχουν φτιάξει δικές τους εκθέσεις. Ε, ήταν πολύ ενδιαφέρον αυτό που ακούσαμε για τις μο... σύγχρονες μορφές επικοινωνίας και τηλεπικοινωνίας αν θέλετε. Ίσως θα πρέπει να χρησιμοποιήσουμε ανεπίσημες μορφές για να ε, επικοινωνήσουμε μεταξύ μας και να κατανοήσουμε καλύτερο ένας τον άλλον. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο πρόσφατα ε, ξεκίνησε το web streaming, δηλαδή να μεταδίδονται στο διαδίκτυο οι διάφορες συνεδριάσεις, ε, αυτό είναι ήδη πάρα πολύ καλό και αυτή η τεχνολογία μπορεί να χρησιμοποιηθεί για το συντονισμό αλλά και οι τηλεδιασκέψεις. Σας ευχαριστώ λοιπόν όλους για τις θέσεις που αναφέρετε, για τη θέση που πήρατε. Είμαστε όπως σας είπα στην αρχή μιας διαδικασίας ε, και σας είπα ποιος είναι ο στόχος μας. Ε, 13.000 παιδιά να ζουν κάθε μέρα να μειώσουμε τον αριθμό των παιδιών που πεθαίνουν κάθε μέρα δηλαδή να υποδιπλασιάσουμε ευχαριστώ πάρα πολύ για τη συμμετοχή σας ε, Ευχαριστώ πολύ κυρία Ζολή στα κοντά στο τέλος της συνεδρίασής μας για τα συμπεράσματα. Έχουμε τη χαρά να έχουμε εδώ τον κύριο Πατ Γκριν, πρόεδρο της ε, Κοινής Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων και Εμπορίου της Ελληνικής Βουλής. Δηλαδή, όπως γνωρίζετε, ασκεί την Προεδρία αυτό το εξάμεινο. Θα σας ακούσουμε λοιπόν και αν έχουμε χρόνο θα έχουμε και συζήτηση. Αν μπορείτε λοιπόν να προφείτε στην διατύπωση των συμπερασμάτων από τις δύο προηγούμενες συζητήσεις. Κύριε Μπριν, παρακαλώ, ε, έχετε 10 λεπτά. Κυρία Πρόεδρε, εξαιρετική η συζήτηση, εξαιρετικά χρήσιμη και πολύ ενδιαφέρουσα. Όλα αυτά να δεικνύουν τον ρόλο μας και την ισχύ που έχουμε όταν μιλούμε με μία φωνή. Το θέμα είναι να επιστρέψουμε όλες τις χώρες μας, τα κοινοβουλιά μας και να φροντίσουμε, να συντονιστούμε και να φροντίσουμε για την συνοχή των προγραμμάτων μας. Να πατήσω φορτιμή στον πρώην συναδελφό μου, τον κύριο Γκέι με τον οποίο συνεργάστηκα επί σειράν ετών. Πρέπει να πω ότι ο Γκέι ε, εργάστηκε σκληρά για τους σκοπούς της ανάπτυξης. Ο εκπρόσωπος της Προεδρίας και του Ιρανικού Κοινοβουλίου ήταν ε, εδώ. Θέλω επίσης να τον χαιρετήσω και να σας πω ότι θα, επιτρέψουμε, θα επιστρέψουμε ε, πιο πλούσιοι στην χώρα μας και στη Βουλή. Πριν λίγο καιρό έλαβε χώρα στην Ιρλανδία, στο Δουβλίνο, η διακοινοβουλευτική διάσκεψη για τα θέματα που συζητούμε και είχαμε την ευκαιρία έτσι να συζητήσουμε όλα τα θέματα. Μια συζήτηση η οποία κατέδειξε ακριβώ τα ωφελήματα τα οποία μπορούμε να πετύχουμε όλοι μα με καλύτερο συντονισμό σε όλου του τομεί. Είναι πολύ ενθαρρυντικό να βλέπουμε εδώ σήμερα το πρωί την ίδια διαδικασία, την ίδια προσπάθεια σε ένα διακοινοβουλευτικό πλαίσιο. Θέλω να συγχαρώ τον μόνιμο συγητή για θέματα συνοχής, ο οποίος ε, καλέσει για καλύτερο προγραμματισμό και συνεργασία. Να ευχαριστήσω και να συγχαρώ την κυρία Ζολή, την οικοδεσπότη μας για τις συστάσεις της. Πολλοί αναφέρθηκαν στην ε, οικονομική κρίση, την παρούσα συγκυρία δηλαδή, τους δημοσιονομικούς περιορισμούς και στην Ευρωπαϊκή Ένωση αλλά και εκτός. Το θέμα λοιπόν είναι επιτακτικό. Να κάνουμε ό,τι μπορούμε για να δούμε πώς δαπανούμε με τον βέλτιστο τρόπο τα δημόσια κονδύλια. Παρά την λιτότητα, και μάλλον λόγω ακριβώ τη λιτότητα. Στην Ιρλανδία Εμεί συνεχίζουμε να αποδίδουμε υψηλή προτεραιότητα στην βοήθεια και αυτό αποτυπώθηκε και σε έρευνα που διεξήγαν διάφορες ΜΚΟ που διαχειρίζονται περίπου 650 εκατομμύρια ευρώ. Η έρευνα αυτή, αυτό το γκάλωπ, έγινε από την TOCUS, μια οργάνωση ομπρέλα ΜΚΟ, που κατέδειξε, επαναλαμβάνω, ότι 76% του πληθυσμού είναι υπέρ των αναπτυξιακών προγραμμάτων. Παρά την κρίση λοιπόν ο κόσμος είναι υπέρ της βοήθειας. Πέραν αυτού, οι φορολογουμένοι θέλουν να ξέρουν πώς δαπανώνται τα κονδύλια αυτά και ότι όντω είναι υποφελία των πραγματικών δικαιούχων. Η υποστήριξη της κοινή γνώμης πρέπει να μας τονώσει ακόμη περισσότερο να μας ενθαρρύνει στις προσπαθίες μας και να προσπαθήσουμε να πετύχουμε περισσότερη συνοχή. Το θέμα δεν είναι μόνο η γεωργία, το κλίμα, οι επενδύσεις κλπ. Οι πολιτικές μας, ας μην ξεχνούμε, μπορούν να έχουν και αρνητικές επιπτώσεις εκτός από τις θετικές στις χώρες δικαιούχους. Η επιδίωξή μας λοιπόν της συνοχής είναι ένα από τα μελήματα. Η κυβέρνηση της Ιρλανδίας είναι προσυλλομένη στην συνοχή. Έχει καταρτήσει και ένα σχετικό έγγραφο. Το 2012 δημιούργησε ένα πλαίσιο για την αηφορική παροχή βοήθειας και φυσικά έχει συμπογράψει και διάφορε συμφωνίε εντό και εκτό Ευρωπαϊκή Ένωση. Υπάρχει μια λευκή βίβλο όπου τονίζεται ότι η συνοχή είναι κάτι παραπάνω από προπόθεση και απέτηση περιορισμού των αρνητικών επιπτώσεων. Είναι η οδός της αηφορίας... και η οδός της επίτευξης των στόχων της Ιρλανδικής βοήθειας. Από το 2006 έχουν γίνει πολλά βεβαίως. Η Ireland 8 ε, περιγράφεται από τον ΟΣΑ και από άλλους διεθνείς οργανισμούς ως πρωταθλητής στην αποτελεσματικότητα της βοήθειας. Μια άλλη έρευνα δείχνει ότι η Ιρλανδία είναι μεταξύ των τριών πιο αποτελεσματικών δωρητών στο top 10 των δωρητών σε όλο τον πλανήτη. Ο οργανισμός Irish Aid είναι ο εθνικός μας οργανισμός παροχής βοήθειας. Τα έχει πάει πολύ καλά. Φυσικά αντιμετωπίζει ακόμη διάφορα προβλήματα και αυτό κατέδειξε και μια έρευνα στην Ιρλανδία όπου τονίζονται οι προκλήσεις που συζητούμε και εδώ σήμερα ιδιαίτερα όσον αφορά τον κατακαιρματισμό και την επικάλυψη των προσπαθειών χωρίς βοηθεία. Πολλοί τόνισαν τον κατακαιρματισμό και την ανάγκη να τον ξεπεράσουμε. Αυτή τη στιγμή πρέπει να μετρήσουμε καταρχήν τον αντίκτυπο των ενεργειών μας. Χρειάζεται να βοηθήσουμε τις χώρες λήπτες με προσωπικό και μέσα. Με την Λευκή Βίβλο επιβεβαιώνουμε την προσήλωσή μας στην ε, ανάπτυξη και τη βοήθεια. Έχουμε καταστρώσει κάποιες διαδικασίες τα τελευταία χρόνια με τις οποίες προσπαθούμε να πετύχουμε περισσότερη συνοχή. Η διακοινοβουλευτική μεικτή επιτροπή εργάζεται για αυτά τα θέματα και προσπαθεί να συγκεράσει την διαθέσιμη τεχνογνωσία για να βελτιώσει τα χαρακτηριστικά της βοηθειάς μας. Η γραμματεία της κυβέρνησης ε, συνομιλεί με διάφορους συμμετέχοντες και την κοινωνία των πολιτών, με ΜΚΙΟ και πανεπιστήμια για το σκοπό αυτό. Επίσης συμμετέχει σε μια άτυπη ανταλλαγή απόψεων για τη συνοχή. Η Air ε, έχει εξοδέψει 30 εκατομμύρια κάθε χρόνο τα τελευταία χρόνια για έρευνα στον τομέα τη βοήθειας. Γίνονται άλλε συναντήσει με θέμα την συνοχή. Υπάρχει ένας άτυπο ε, μηχανισμός συνεργασία και συντονισμού με γνώμονα τον εξορθολογισμό της προσπαθειάς μας. Αυτό είναι πολύ σημαντικό. Αυτή η προσπάθεια αφορά όλα τα Υπουργεία, όλους τους ε, κυβερνητικούς ε, φορείς. Πέρσι, η Κοινοβουλευτική Επιτροπή για τις Εξωτερικές Σχέσεις και το Εμπόριο, της οποίας προεδρεύω, τόνισε την ανάγκη συνοχής μεταξύ της Ιρλανδικής βοήθειας και της γενικότερης πολιτικής της κυβέρνησης. Ο Μάλκομ Μπρούς ε, το θύμισε αυτό λίγο νωρίτερα είπε ότι υπάρχει ε, σχέση και σύνδεση μεταξύ εμπορίου και πολιτικής στον τομέα της ε, βοηθείας. Οι πρεσβείς μας στην Αφρική είναι υποχρεωμένες να αναφέρουν τη σχετική πρόοδο κάθε χρόνο που γίνεται στον τομέα. Η Επιτροπή μα επίση, αλλά και άλλε επιτροπέ, συνεργάζονται με την Irish ε, Aid με στόχο την διαφάνεια και την καταγραφή των αποτελεσμάτων. Ο συνάδελφος από το Βέλγιο το είπε πολύ σωστά προηγουμένως ότι τα κοινοβούλια πρέπει να επιβλέπουν, να επιτηρούν την κατάσταση. Οι βουλευτές, κάθε καθένας στη χώρα του, πρέπει να γνωρίζουν ενώ για τις χώρες ε, λήπτες, πόση βοήθεια και ποια βοήθεια έχετε από ποια χώρα. Για να έχουν ένα ρόλο ε, επιβλέψης και επιτηρήσεως, τα κονδύλια να πηγαίνουν εκεί που πρέπει. Επίσης ζητούμε η κυβέρνηση να στέλνει πιο καθαρά το μήνυμα για την αποτελεσματικότητα της βοήθειας. Η κυβέρνηση λοιπόν υποστηρίζει μεταξύ άλλων και την καλή συνεργασία με τις ΜΚΟ. Είναι κάτι το οποίο νομίζω σας βρίσκει όλους σύμφωνος απαιτείται συντονισμό των δωρητών για να αποφύγουμε επικαλύψει και να είμαστε πιο αποτελεσματικοί. Η αρχή αυτή εκφράζεται και σε επίπεδο Ευρωπαϊκή Ένωση. Η Ευρωπαϊκή Ένωση έλεγε δεσμεύσει εν προκειμένου όσον αφορά την αποτελεσματικότητα των προγραμμάτων βοήθεια. Όπω γνωρίζετε, τον Μάιο του 2012 η Επιτροπή και η WAS αποφάσισαν να έναν κοινό προγραμματισμό. Στα τέλη του 12 επελέγει η Αιθιοπία ως ε, παράδειγμα, ως ε, πιλωτικό πρόγραμμα για τον κοινό προγραμματισμό. Έχουμε πλέον ε, θετικά σημάδια από αυτόν τον κοινό προγραμματισμό στην Αιθιοπία και αυτό θα ενθαρρύνει τον συντονισμό της καλύτερης διακυβέρνησης και των τομεακών προγραμμάτων. Η Ιρανική Πρεσβεία στην Αντίσσα που επισκέφθηκε πέρσι, διαδραματίζει πολύ σημαντικό ρόλο στον κοινό προγραμματισμό. Προσβλέπουμε στην ολοκλήρωση του συγκεκριμένου έργου που θα αποδείξει την αξία του κοινού προγραμματισμού στην Αιθιοπία. Θα υπογράψουμε την κοινή στρατηγική τις επόμενες εβδομάδες. Ελπίζω ότι το σχέδιο αυτό στρατηγική θα πετύχει για να υλοποιήσουμε ένα κοινό όραμα αντιμετώπιση των κοινών οραμάτων για την ανάπτυξη και τη βοήθεια. Και ελπίζω ότι η γενικότερη αυτή στρατηγική θα ενταχθεί σε μια γενικότερη στρατηγική της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και πρόεδρε, η Επιτροπή μου, η Επιτροπή Εξωτερικών Σχέσεων πήγε στην Freetown, στη Σιέρα Λεόνι, για να δούμε τι κάνουν εκεί οι Ιρλανδοί και τι κάνει το Γραφείο Ιρλανδικής Βοηθεία. Και εντυπωσιάστηκα πρέπει να πω από τον τρόπο με τον οποίο μια μικρή ομάδα συνεργάζεται με τοπικούς και διεθνείς φορείς για τα επιστημιστικά προγράμματα, για τα προγράμματα αγροτικής ανάπτυξης, για προγράμματα στον τομέα της υγείας. Ο συντονισμός των δωρητών προκειμένου σε μια τοπική κλίμακα βεβαίως έδειξε πόσα πλεονεκτήματα έχει και είμαι σίγουρος ότι και άλλες επιτροπές το έχουν δει στα δικά τους προγράμματα. Όλα αυτά τόνισαν για άλλη μια φορά την αξία του συντονισμού μεταξύ δωρητών να βοηθήσουμε χώρε όπου η παιδική θνησιμότητα θερίζει. Και αυτό συμβαίνει και σε άλλε βεβαίω χώρε. Έχουμε σεξουαλική βία, υποανάπτυξη και άλλα προβλήματα που πρέπει να αντιμετωπίσουμε. Να εντείνουμε λοιπόν τι προσπαθίε μα μαζί με τα άλλα κοινοβούλια και να κοιτάξουμε να κάνουμε κάτι για του ανθρώπου των οποίων οι ζωέ εξαρτώνται από τι δικέ μα αποφάσει. Κύριε Πρόεδρε, κλείνω λέγοντα ότι σα φίλω ευχαριστίε για την διοργάνωση αυτής της ε, συνεδρίασης που έφερε κοντά το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και τα Εθνικά Κοινοβούλια. Θα φύγουμε έτσι πλουσιότεροι και θα ασκήσουμε πίεση στις κυβερνήσεις μας για να ελοπίσουμε τις συστάσεις σας. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ. Τώρα έχουμε κάποια λεπτά στη διάθεσή μας ε, για μια ανταλλαγή απόψεων με τον ε, πρόεδρο της ε, Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων και Εμπορίου του Ιρλανδικού Κοινοβουλίου. Όσοι παρούν το λόγο όμως παρακαλώ να περιοριστούν στο ένα λεπτό. Αν δεν ε, επιθυμείτε να πάρετε το λόγο, ευχαριστώ τον πρόεδρο της Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων για την ε, συνεισφορά του. Ευχαριστώ όλους όσους συμμετείχαν σε αυτή τη συνεδρίαση για τον πλούτο των απόψεων που ακούστηκαν ε, σήμερα το πρωί και για τα θέματα που συζητήσαμε. Φυσικά πρέπει να εργαστούμε περαιτέρω για να πετύχουμε τη συνοχή της αναπτυξιακής πολιτικής και όπως είπα και εισαγωγικά η συνοχή της αναπτυξιακής πολιτικής δεν ε, είναι απλώς ε, κάτι μεταξύ κρατών μελών και κοινοβουλίων, πρέπει να το σκεφτούμε το όλο ζήτημα καθολικά και οι παράνομες ε, χρηματοοικονομικές ροές ε, που ε, εγκαταλείπουν τις αντισόμενες χώρες είναι 10 φορές μεγαλύτερες από την απταξική βοηθεία που τους παρέχουμε. Έτσι λοιπόν και τα δικά μας φορολογικά καθεστώτα συνεισφέρουν τα μέλη στην κατάσταση χρηματοδότησης των αναπτυσσόμενων χωρών και αυτό είναι ένα θέμα που θα πρέπει να εξετάσετε στις αντίστοιχες χώρες σας. Ολοκληρώνουμε τώρα τη συνεδρίαση αυτή και σας καλώ όλους να ε, συμμετάσχετε εδώ σε ένα ελαφρύ γεύμα που θα σερβιριστεί έξω από το ημικύκλιο και μπορούμε να συνεχίσουμε με την ε, ανταλλαγή των απόψεών μας ε, με ένα ποτήρι κρασί. Σας ευχαριστώ όλους.